Good morning again. Καλή σας μέρα και πάλι. Καλημέρα σας. Colleagues, dear, let's proceed. Let's proceed. We had a coordinators meeting. Ας αρχίσουμε. Ε, έγινε η... Points number nine. Ε, κάναμε τη συνάντηση των συντονιστών και τώρα προχωρούμε με τις συνεδρίες Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και έχουμε στην ατζέντα δύο ψηφοφορίες. Πρώτη ερώτηση, την ηλεκτρονική σας κάρτα τη φέρατε για να κά Κυρία Μακομπέη δεν έχετε Συγγνώμη δεν την έφερα Θα σηκώ το χέρι μου Άρα λέει ο πρόεδρος διανατάσεως της χειρός ψηφοφορίας. Η κυρία Μακοβέη δεν έχει την κάρτα της. Λοιπόν, στο σημείο 7, ε, το σημείο 9 είναι η θέσπιση ενό μηχανισμού αξιολόγηση για την επαλήθευση εφαρμογή του κεκτημένου του Σέγγεν. Εισηγητή ο κ. Κοέλο, θέλετε το λόγο. Όχι, πρόεδρε, αφού το συζητήσαμε χτε, πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. ο εισηγητής προτείνει να απορριφθεί η πρόταση της Κομισιόν. Επ' αυτού ψηφίζουμε λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ της απόρριψης της πρότασης της Κομισιόν. Α, όχι, να αρχίσουμε ανάποδα. Λοιπόν, ποιος Ποιος ψηφίζει κατά του κειμένου της Κομισιόν. Μεγάλη πλειοψηφία, οπότε ακολουθούμε την πρόταση του εισηγητή. Μετά, στο σημείο 10 έχουμε το μηχανισμό αξιολόγηση για την παλήθευση εφαρμογή του κεκτημένου του Σέγγεν. Το ίδιο. Ποιος ψηφίζει κατά του κειμένου της Κομισιόν ή μάλλον ή υπέρ του εισηγητή. κατά υπέρ του κειμένου της Κομισιόν προφανώς ουδής άρα απορρίπτεται η πρόταση Κομισιόν υποστηρίζουμε τον εισηγητή Προχωρούμε τώρα στο σημείο 11 για τον οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και μετά λειτουργική διαχείριση συστημάτων SIS2 και VIS. Λοιπόν, ο εισηγητής και για τα δύο θέματα είναι ο κ. Κάρλος Έχετε το λόγο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι μεγάλη ευχαριστήσή μας ε, με την ε, πρωτοβουλία αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπενθυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές ζήτησε την ρύθμιση αυτού του θέματος και το γεγονός ότι παρουσιάζει πλέον το κείμενο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημαίνει ότι έτεινε ευήκον ούσο προς τις ε, εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων θα ήθελα να αναφέρω κάποια στοιχεία. Πρώτον, θα ήθελα να πω ότι όπως κάναμε σε παρόμοιες ε, διαδικασίες και στον, στο πλαίσιο του σεβασμού των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου δεν έχει νόημα να έχουμε διαφορετικές νομοθετικές διαδικασίες εφόσον πρόκειται για το ίδιο αντικείμενο. Κατά συνέπεια η προσέγγιση μας θα αποτελέσει μια συνολική αντιμετώπιση ως δέσμη, ως πακέτο όπως λέμε. Έτσι λοιπόν θα αναλύσουμε τα θέματα αυτά ως δέσμη. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, αναφέρθηκε από κάποια κράτη-μέλη η ιδέα ότι οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να δοθούν σε μια υφιστάμενη ήδη υπηρεσία. Θα ήθελα να πω ότι κατά την απόψή μου αυτή είναι μια λάθος λύση. Θα πρέπει να έχουμε μια υπηρεσία ειδική για τα θέματα που αφορούν την πληροφορική. Τα θέματα αυτά να δοθεί η αρμοδιότητα στο Frontex ή στην Europol αντιβαίνει με αυτή την ιδέα που μόλις παρουσίασα. Διότι δεν διαχειρίζεται μόνο, αλλά ωφελείται, καταναλώνει ούτως υπήν και τα δεδομένα που επεξεργάζεται. Το δε επιχείρημα του κόστους δεν νομίζω ότι είναι συναφές το ένατο κεφάλαιο της αξιολόγησης αντικτύπου αναφέρει ότι η δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας ε, επισύρει ουσιαστικά το ίδιο κόστος με το αν αποδοθεί η αρμοδιότητα αυτή σε υφιστάμενη υπηρεσία. Οπότε το κόστος, η δαπάνη δεν είναι κέριο επιχείρημα. Σε ό,τι αφορά την ουσία. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλές εξειδικευμένες, ε, μάλλον προσπάθεια εξειδίκευσης των προτάσεων που είναι γενικές σε ό,τι αφορά τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας αλλά και τον ρόλο που θα έχει αυτή η υπηρεσία σχετικά με μελλοντικά ενδεχομένω συστήματα ή για το θέμα για το ποιος είναι ο κάτοχος, ο κύριος των δεδομένων. Από αυτή την άποψη πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρό η έγκριση μιας ε, νομικής βάσεως για την διαχείριση αυτού του συστήματος δεν μπορεί να λάβει μορφή λευκής επιταγής. Δηλαδή έναν κανόνα ο οποίος θα επιτρέπει στο ίδιο καλάθι να βάλουμε τα πάντα. Χωρίς τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει λοιπόν πολλή δουλειά για την βελτίωση του καθεστώτος προστασίας ε, των δεδομένων. Το άρθρο 25 περιλαμβάνει απλώς μια γενική, έναν γενικό κανόνα με το άρθρο 45 του κανονισμού 2001 και νομίζω ότι πρέπει να βελτιωθεί. Και από αυτού αναμένω με πολλές προσδοκίες την έκθεση που υποβάλαμε στον Ευρωπαϊκό ε, διαμεσολαβητή για την προστασία των δεδομένων. Τώρα, η πρόταση αναφέρει την ε, ύπαρξη ενός ε, βιομετρικού συστήματος το οποίο θα είναι διαθέσιμο και για το σύστημα VIS αλλά το οποίο θα διευρυνθεί σε μια περαιτέρω φάση στο SIS2 και στην Eurodac. Υπάρχουν πολλά θέματα που τίθενται εδώ δημιουργούμε μια τεράστια βάση δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων στην Ευρώπη. Και υπάρχουν και θέματα που θα προκύψουν στο μέλλον, το exit system ή το electronic travel authorization. Τέλος, για να ολοκληρώσω, Πρόεδρε, στην πρώτη μου αυτή τοποθέτηση, το Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί αγαστά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, όπως κάνουμε πάντα και όπως κάναμε για όλα τα νομοθετικά μέσα στα πλαίσια του ΣΥΣ, ούτως ώστε να καταλήξουμε στη συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Αν εργαστούμε αποτελεσματικά και επιτύχουμε την άμβλυνση των διαφορών μας, δεν αποκλείω να καταλήξουμε σε συμφωνία και σε πρώτη ανάγνωση. Και πιστεύω ότι είναι και η ώρα τώρα, Πρόεδρε, αν συμφωνείτε, να ακούσουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου στα πλαίσια της πρώτης αυτής ανταλλαγής απόψεων που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο ή η εκπρόσωπος της Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής αυτή και τον εισηγητή για όλα αυτά που είπε με τα οποία συμφωνούμε απόλυτα. Τα περισσότερα επιχειρήματα που ανέφερε ο εισηγητής θα ήταν και τα δικά μας επιχειρήματα. Θα ήθελα επίσης να εκ μέρους του κυρίου Μπαρόσα ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορούσε να έρθει σήμερα γιατί θα, ήταν, θα ήθελε να παραστεί και αυτό στη συζήτηση αυτή αλλά είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Οι δέσμοι αυτή καθεαυτή που προτείνεται και που όπως είπε και ο εισηγητής είναι μια δέσμη που περιλαμβάνει τον κανονισμό και την ε, ε, απόφαση και το δημοσιονομικό δελτίο και τα λοιπά. Ε, εδώ να έχω μια παρένθεση και λέω ότι τα, καλά τα νέα από την Ιρλανδία που είχαμε τούτη εβδομάδα ήταν, ε, επηρεάζουν ιδιαίτερα την κατάσταση γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας αλλάζει ορισμένα πράγματα ο κανονισμός βέβαια συνεχίζει να ισχύει αλλά η απόφαση πρέπει να αλλάξει να επανυποβληθεί βάσει του άρθρου 87 της συνθήκης λοιπόν ε, η διαδικασία της συναπόφασης επίσης εφαρμόζεται εδώ και αυτό νομίζω ότι θα διευκολύνουν την ε, υιοθέτηση της ε, ε, δέσμης αυτής. Τώρα, με δύο λόγια για την όλη λογιστική. Ακούσαμε από τον εισηγητή ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι γιατί φτιάχτηκε η πρόταση αυτή. Βεβαίως... Ε, υπάρχει κοινή δήλωση πριν από δύο χρόνια όπου όλα τα, όλοι τα θεσμικά όργανα εξέφρασαν τη βούλησή τους. Υπάρχουν και νομοθετικές πράξεις για όλα τα εφιστάμενα συστήματα και για το Eurodac και ε, από εκεί και πέρα ε, έχουμε κατά νου ότι και μια διαχειριστική αρχή, μια agency της Κομισιόν θα πρέπει να αναλάβει τη διαχείριση όλων αυτών τα επιχειρήματα για αυτή την κανονιστική αρχή, ε, την κανονιστική υπηρεσία, την agency, παρουσιάστηκαν από τον ο, εισηγητή, αλλά για τη διακυβέρνηση αυτού του οργάνου, για τη διοίκηση αυτή τη agency, να πω ότι βεβαίω η διοίκηση αυτή, ε, τα διοικητικά θέματα, ε, διοικητική δομή θα είναι όπως και των άλλων υπηρεσιών, ε, διοικητικό συμβούλιο, διευθυντή, και από εκεί και πέρα ε, το μόνο που θα είναι διαφορετικό από τις άλλες agencies είναι ότι θα υπάρχουν και συμβουλευτικές ομάδες. Γιατί, διότι κάθε ένα από τα συστήματα που θα καλύπτονται από αυτή την υπηρεσία, από αυτό το γραφείο, απαιτούν γνώσεις ειδικέ που ενδεχομένως να μην έχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι αν είχαμε συμβουλευτικές ομάδες μια για την κάθε μια από, το κάθε ένα από τα συστήματα θα βοηθούσαμε και τη δουλειά του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτά λοιπόν για τη διοίκηση τη agency αυτή. Ε, κατά τα άλλα είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω ρωτή σχετικά αν θέλετε. Τώρα προχωρώ. The ε, presentation ε, of... Α, προχωρώ στο κόστος και τα θέματα αυτά τα ανέφερε ο κύριος Κοέλο βεβαίως ε, απλώ επαναλαμβάνω και επιβεβαιώνω ότι εκτίμηση που κάναμε ε, συνέκρινε το κόστος της, του βασικού συστήματος θέλετε όπως είναι αυτό το SIS όπου τρέχουν διαχειρίζονται τα συστήματα τα κράτη-μέλη και με το κόστος που θα είχε η διαχείριση από μια agency υπάρχει και μια τρίτη εναλλακτική ε, που βλέπετε στο κείμενό σας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, από την σύγκριση αυτή που κάναμε είδαμε ότι δεν θα γίνονταν οικονομίες με το να δώσουμε τη διαχείριση σε μία από τις υφιστάμενες υπηρεσίες, από τα υφιστάμενα γραφεία. Διότι σε πρώτη φάση ε, το κόστος ε, της διαχείρισης θα ήταν το ίδιο για μια υφιστάμενη agency, μια καινούρια agency ενώ η δημιουργία μιας ειδική καινούρια agency μακρόχρονα θα είχε ωφέλη. Ο εισηγητής ανέφερε όσον αφορά τους στόχους ε, ότι δεν φαίνονται σαφώς οι στόχοι στο κείμενο που έχουμε φτιάξει και η σχέση των τωρινών αν μπορούμε να πούμε στόχων με τους μελλοντικού στόχους για την επέκταση των συστημάτων ασφάλεια ε, εσωτερική ασφάλεια κλπ. Ναι, ήταν συνειδητό αυτό επιλέξαμε να αναφερθούμε απλώς στη νομική βάση του κάθε από τα συστήματα που καλύπτονται διότι φανταστήκαμε ότι αυτό μας έδινε μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη κατανόηση των το αυτόν που επιδιώκουμε και για το ΣΥΣ2 και για το ΒΙΣ και για το Eurodac ε, υπάρχουν ε, στόχοι για το κάθε σύστημα εν λεπτομέρειες το να προσπαθήσουμε λοιπόν αυτούς τους επιμέρους στόχους του κάθε ενός συστήματος να τους βάλουμε μαζί σε ένα κείμενο θεωρήσαμε ότι δεν θα ήταν καλό βεβαίως μπορούμε να επανεξετάσουμε το ζήτημα αν θέλετε και να κάνουμε σαφέστερη την πρόταση τώρα για το μέλλον το κείμενο φτιάχτηκε με τέτοιο τρόπο τους ώστε να επιτρέπει την επέκταση αν θέλετε αν υπάρχουν αν παρθούν πολιτικές αποφάσεις για νέες νομοθετικές πράξεις, για νέα μεγάλα συστήματα πληροφορικής ε, στην Ευρώπη κτλ. Όλα αυτά μπορούν να προσθεθούν και ε, μπορούμε, μπορεί να επεκταθεί η πρόταση. Είναι Βεβαίω κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε αν και εφόσον πάρθει η πολιτική απόφαση. Τώρα για την προστασία των δεδομένων είναι προφανώς κάτι, ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ότι ε, σας ανησυχεί. Στο άρθρο 25 αναφερόμαστε στην στον υφιστάμενο κανονισμό για την προστασία των δεδομένων και για τους... Τότε όταν κουβεντιάζαμε και τους στόχους ε, σκεφτήκαμε ότι η agency η καινούρια αυτή θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες ελέγχου για την προστασία των δεδομένων πλήρως. Οι σχετικές αρμοδιότητες υπάρχουν, οι DPS και τα λοιπά ελέγχη πισκέψεις επισκέψεις επιτόπου κτλ. Όλα αυτά πρέπει να τηρούνται και θα πρέπει να υπάρχει και ένα άτομο ή ένας ε, αξιωματικούς ειδικά για τους ελέγχους που να εργάζεται στην agency και να ασχολείται με το θέμα αυτό. Τώρα για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το αναφέρεται αυτό στο κείμενο ε, πρόκειται για μια agency του πρώτου πυλώνα και βεβαίως ε, από αυτό απορρέουν και οι σχετικοί έλεγχοι και αρμοδιότητες. Επιπελέον το κείμενό μας λέει ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι ενισχυμένος ε, για οποιαδήποτε, σε σχέση με οποιαδήποτε αλλαγή ε, ενημερώνεται το κοινοβούλιο δηλαδή για οποιαδήποτε ε, αλλαγή ε, που η οποία μπορεί να έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο και, μετά διαβιβάζει το κοινοβούλιο μέσα στους κομισιόν. Είμαι στη διάθεση σας για ερωτήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάμαστε εκ μέρους της Προεδρίας του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ για τη μελλοντική μας συνεργασία με το Κοινοβούλιο για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τόμας Κοέλιο, τον εισηγητή, για την εξαιρετική παρουσίασή του. Επίσης ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί και η δική της παρουσίαση ήταν εξαιρετική. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και πιστεύουμε ότι θα μας επιτρέψει να κάνουμε προόδους το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει συνένεση για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να χειριστούμε αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται μια παρουσίαση αυτή τη στιγμή για το πώς θέλουμε εμείς να χειριστούμε τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο, ε, αλλά ευχαρίστως να απαντήσω σε οποιασδήποτε ερωτήσεις σας. Ποιος θα ήθελε το λόγο, ο κύριος Άλβαρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι και εγώ εκ μέρου τη πολιτική μου ομάδα που συζητάμε αυτό το θέμα και με μεγάλη χαρά συνεργαζόμαστε με τον ε, κύριο Κοέλιο. Ε, ξέρουμε ότι και το ΕΛΚ έχει στείλει ένα πολύ αξιόλογο εισηγητή που θα χειριστεί με μεγάλη επιδεξιότητα αυτό το θέμα. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις ε, πριν ε, εξετάσουμε λεπτομερώς το έγγραφο, χωρίς ε, να επαναλαμβάνω βέβαια αυτά τα οποία ήδη είπε ο συνάδελφος κ. Κοέλιο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση για δημιουργία ενό οργανισμού, μιας agency, για να δούμε κατά πόσο είναι ρεαλιστικό και εφικτό. Είναι κάτι το οποίο προβλέπεται να εφαρμοστεί το 2012 ε, συμπεριλαμβάνοντα ε, ε, το ΣΥΣ2. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί το ΣΥΣ2 μέχρι το 2012. Και ελπίζω να όντω να συμβεί αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και χωρίς να θέλουμε να κατηγορήσουμε την Επιτροπή για τη μη λειτουργία μέχρι τώρα, αλλά πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να έχουμε τη διαχείριση από έναν οργανισμό και να δούμε αν ε, θα συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα και οι βάσει δεδομένων που ήδη υπάρχουν ε, στα υπάρχοντα συστήματα όπως το SIS ε, και το VIS. Για την προστασία δεδομένων, ήδη ανέφερε ο κ. Σκοέλιο, στο άρθρο 25 μιλάμε για το θέμα αυτό, αλλά αυτό είναι το σωστό άρθρο, μιλάμε για, για μια ρύθμιση του πρώτου πυλώνα Φαίνεται ότι πρόκειται για ένα οργανισμό του πρώτου πυλώνα και στην αιτιολογική σκέψη 10 ε, μιλάμε για τον, ε, αναφέρει το τίτλος 4 τα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ε, και δεδομένα που υπάρχουν στον τίτλο 4. Δηλαδή υπάρχει μια ρήτρα που αφήνει ε, ανοιχτό πεδίο για τη διαχείριση από ένα κεντρικό οργανισμό, για τη διαχείριση των δεδομένων από ένα κεντρικό οργανισμό. Δεν ξέρω αν υπάρχει μικρότερη ευελιξία. και θα πρέπει να, να δούμε κατά πόσο θα μπορεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να δούμε ποιες βάσεις δεδομένων μπορούν να συμπεριλαμβάνονται. και θα ήταν πραγματικά χρήσιμο σημαντικά σημεία όπως η πρόσβαση η ανταλλαγή δεδομένων ε, μεταξύ κρατών μελών ε, να μπορούν να ρυθμιστούν σαφώς και θα πρέπει να γίνεται και παραπομπή στους ισχύοντες κανονισμούς για το SIS, το VIS και το Eurodac ούτως ώστε ε, ένας αρμόδιος οργανισμός ε, να μπορεί να ε, χρησιμοποιεί αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν για, αυτούς, για αυτά τα συστήματα. Στον τύπο διάβασα ότι δέχεται αυτός ο οργανισμός να δημιουργηθεί και στην Ισλανδία. Και πιστεύω ότι επειδή ακριβώς χειρίζεται ευαίσθητα δεδομένα που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν και ποινικά στοιχεία, θα πρέπει να δημιουργηθεί μέσα σε μία δομή ε, ώστε να αποτρέπεται ακόμη και ο πειρασμός ε, κατάχρησης των δεδομένων. μπορεί να τρέχω μεγάλη συμπάθεια για την Ισλανδία, αλλά αναρωτιέμαι αν επελέγει η Ισλανδία ως πιθανός ε, τόπος εγκατάστασης, γιατί έχει ήδη η Ισλανδία μεγάλη πείρα για την ε, διαχείριση δεδομένων ε, και αν πιστεύετε ότι θα είναι σκόπιμο να επιλεγεί ως τόπος αυτού του οργανισμού η Ισλανδία. για το ε, προπολογισμό των 130 εκατομμυρίων ευρώ νομίζω ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε και μέχρι ε, το 2012 να το εξετάσουμε, να δούμε πόσοι ε, συνεργάτες θα χρειάζονται, αν χρειάζονται 120, αν θα χρειάζονται μόνο 50 άτομα προσωπικό. Είναι ήδη μεγάλη η αριθμή των ατόμων που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ε, η αιτιολογική σκέψη 10 ε, έχει μια αναφορά που συμπεριλαμβάνει και την ε, μνήμα άλλων υφισταμένων ζητημάτων. Υπάρχει και το σύστημα της συνθήκης του, του και πρέπει να δούμε αν μέσα στο πλαίσιο αυτού του οργανισμού θα πρέπει να συγκεντρωθούν οι βάσεις δεδομένων και αν θα γίνεται ε, η διαχείριση μέσω αυτού του οργανισμού ε, ή αν θα ε, συνδυάζει τις δραστηριότητες των υφισταμένων οργάνων για να χειριστεί αυτά τα θέματα, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες διασυνδέσεις. Και υπάρχει και ένα σχετικό κείμενο της Επιτροπής για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων. ώστε να και ο ε, και η απέτηση για την αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα του οργανισμού. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς θα λειτουργήσει αυτός ο οργανισμός. Ε, και να συζητήσουμε ε, και το άρθρο 26 για άλλες σχετικές πληροφορίες και το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Ε, ε, πιστεύω ότι μιλάμε για το πεδίο της συναπόφασης και ούτως ή άλλως δεν θα έχει γίνει ματέως η δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα και με τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Πάντως χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνεργασία που θα έχουμε με τον συνάδελφο κ. Κοέλιο να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Αλεξάνδρου Άλβαρο νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε και να εξετάσουμε κατά πόσο το μέτρο αυτό είναι ε, απαραίτητο και για ποιο λόγο θα ήθελα να έχω μια σαφέστερη αν θέλετε εικόνα των στόχων και τις ανάγκες που οδήγησε στη, που στη δημιουργία ενός νέου οργανισμού τα στο μέτρο αυτό η προστασία των δεδομένων ε, μπαίνει σε δεύτερο πλάνο αυτό δεν με ικανοποιεί και θα πρέπει λοιπόν να το προσέξουμε αυτό και θα πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε βασικές αρχές που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων. Τι σημαίνουν εδώ οι οικονομίες αν θέλετε ε, δημιουργία συνεχώς νέων θέσεων, νέων τραπεζών δεδομένων οι οποίες όμως μελλοντικά συγχωνεύονται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο λοιπόν εδώ θα πρέπει να θέσει πολύ συγκεκριμένα όρια διότι το να πει απλώς ότι δεν πρόκειται να συλλεχθούν και να ε, συνδυαστούν και να διαδοθούν ε, δεδομένα εδώ είναι ε, ωραία λόγια αλλά επί ε, για μένα οι τράπεζες δεδομένων έχουν κάποιο πρόβλημα γιατί σε ε, ή οποιοδήποτε συνδυασμός δεδομένων σημαίνει και νέα συλλογή στοιχείων και νέα επεξεργασία και άλλες μεθόδους ε, διάδοσης. να σας πω ένα παράδειγμα. Το Eurodac παίρνει ε, δακτυλικά αποτυπώματα από όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζητούν εδώ, να, ε, που ζητούν στην Ευρώπη άσυλο η συλλογή των στοιχείων αυτών και ο συνδυασμός τους με τα στοιχεία του Σέγγεν ή με τα στοιχεία του, του Βίζ για τις ε, θεωρήσεις ε, δημιουργεί ένα κρυκτικό μείγμα δεδομένων και τελ, ε, ο συνδυασμό αυτών των στοιχείων μου δημιουργεί ένα πρόβλημα ότι θα υπάρχει μια καινούργια agency ολόκληρη που θα ασχολείται με αυτά τα πράγματα οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ αυστηρό με τα δεδομένα αυτά η... πρέπει να ζητεί στοιχεία για το τι θα γίνουν τα δεδομένα που συλλέγονται πριν από τη συλλαγή τους όχι να συλλέγονται πρώτα τα στοιχεία και μετά να δημιουργούν να χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς πέραν αυτού για τον οποίο συνελέγησαν Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ και εμείς αντίστοιχες αμφιβολίες έχουμε όπως ο προλαλής γιατί χρειάζεται να φτιαχτεί πρώτα πρώτα ένας κανονιστικός οργανισμός, μια κανονιστική agency για αυτή τη δουλειά. Διότι εδώ μιλάμε για μια, ένα οργανισμό που θα διαχειρίζεται ένα μονοπόλιο δεδομένων ο, ουσιαστικά. Και εδώ ε, στο, στα πρώτα άρθρα άλλωστε του κανονισμού συνεχώς αναφέρεται ο, και άλλων μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων και άλλων μεγάλων συστημάτων και στο άρθρο 6 συγκεκριμένα αναφέρονται και πιλωτικά προγράμματα τα οποία μπορεί να ε, ε, με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί η agency αυτή. Εγώ δεν μπορώ να δώσω λευκή επιταγή για την ε, διαχείριση οποιοδήποτε μεγάλου πληροφοριακού συστήματος ή πιλωτικού προγράμματος στην, στον οργανισμό αυτό. Γιατί δημιουργούμε ένα τέτοιο μονοπόλιο. Πρώτη ερώτηση αυτή. Δεύτερη. για την αναγκαιότητα της ε, agency αυτής. Δεύτερο ερώτημα τώρα για την προστασία των δεδομένων. Δεν βλέπω να λέγονται εδώ πολλά πράγματα για την προστασία των δεδομένων. Είναι ένιγμα για μένα πως ε, τι προστασία προβλέπεται. Εγώ λέω ναι βεβαίω να υπάρχει ένας υπάλληλο ε, ειδικό για τον έλεγχο, για την προστασία των δεδομένων, αλλά υπάρχει κι άλλο ένα ερώτημα. Κατά τα άλλα η agency πώς ελέγχεται. Εμείς σαν κοινοβούλιο, σαν ευρωβουλευτές τι δυνατότητες έχουμε να ελέγξουμε αυτό το, το καινούριο μολόχ, το καινούριο μονοπόλιο που δημιουργούμε. Για να μην σας πω ότι προφανώς και ο πολίτης δεν έχει κανένα, ε, καμιά τέτοια δυνατότητα, αυτή δεν την έχουμε εμείς κατά μείζωνα λόγο βεβαίως. Άρα κάτι πρέπει να, που, να σκεφτούμε σχετικά και κάποιος ε, είπε προηγουμένως ότι πρέπει να ε, ότι επειδή εδώ πρόκειται για καυτά θέματα θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο την πρόταση και όντως νομίζω ότι πρέπει να μελετηθεί πολύ περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Στάνοκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και θα ήθελα καταρχήν εκ μέρου τη ομάδα μου να συγχαρώ τον κύριο Κοέλιο και να εκφράσω την ικανοποίησή μα για το γεγονό ότι είναι εκείνο ο εισηγητής. Είμαστε πεπισμένοι ότι έχει επαρκή εμπειρία και με χαρά θα συνεργαστούμε μαζί του. Η θέση επαναλαμβάνω τη θέση των, της ομάδας μου των Πρασίνων ε, σχετικά με τη χρήση βιομετρικών στοιχείων. Γνωρίζουμε το πώς έχει η κατάσταση για τη χρήση βιομετρικών στοιχείων για τις θεωρήσεις διαβατηρίου σε σχέση με αυτή τη βάση δεδομένων και τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τον νέο οργανισμό. Θα ήθελα μια απάντηση από την Επιτροπή για τον τόπο που θα φιλοξενηθεί αυτός ο νέος ε, οργανισμός. Μας ενδιαφέρει το θέμα των κινδύνων που έχουν σχέση με την προστασία δεδομένων. Και η θέση μας, όπως και του εισηγητού, είναι να περιμένουμε κάποια γνωμοδότηση από τον ε, επόπτη προστασία δεδομένων και να συνεχίσουμε τη συζήτηση μετά από αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριος Δίας Δεμέρας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις ικανότητες του Κάρλος Κοέλιο για την σύνταξη μιας τέτοιας εκθέσεως τόσο πολύπλοκης και ευαίσθητης. Δεν μίλησα ούτε με τον Κάρλος ούτε με την ομάδα του, θα το κάνω. Ήθελα απλώς εδώ να αναφέρω κάποιες αμφιβολίες που εκφράστηκαν Πόλικό ημερικός από κάποιους ε, συναδέλφους που μίλησαν πριν από μένα. Συμφωνώ με κάποιες από τις ιδέες που παρουσίασε ο Αλεξάνδρ Άλβαρο πιο συγκεκριμένα. Πάντως έχω ένα ερώτημα, όχι προς τον ε, ε προς την Κομισιόν, αλλά κυρίως προς το Συμβούλιο που ζήτησε την άποψή μας. Εκουσίως δεν είναι λεπτομερείς οι διατάξεις. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν να είναι. Η ενσωμάτωση μελλοντικών συστημάτων στην υπηρεσία. Ένα διοικητικό συμβούλιο εξειδικευμένο για να ξέρει γιατί μιλάει. Ιδάλλως θα προκύψει πύργος της Βαβέλ ΣΥΣ, ΒΙΣ, Eurodac. Κλεμμένα αυτοκίνητα, αγνοούμενοι, παραχάραξη του ευρώ, παιδοφιλία, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, τρομοκρατία, δίκτυα, ε, ε, εργαστήρια ε, αστυνομικής ε, ε, φύσεως όλα αυτά να ενσωματωθούν είναι αδύνατον και λέγω αδύνατον εκ Το πρώτο που πρέπει να γίνει λοιπόν και θα μιλήσω με την πολιτική μου ομάδα είναι να περιορίσουμε το εύρος τη φιλοδοξία των στόχων που θα έχει μια τέτοιου είδου υπηρεσία για τη διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής στον τομέα μάλιστα της ε, ασφάλειας, ε, δικαιοσύνης και ελευθερίας. Θέτω λοιπόν το ερώτημα στην Κομισιόν, αλλά κυρίως στο Συμβούλιο. Ο κύριος Μπουζουτήλ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον Κάρλος για τη δουλειά που έχει κάνει για το θέμα αυτό. Πάντοτε έχω την εντύπωση όταν μιλάμε για τα εξωτερικά σύνορα και το Σέγγεν, πάντοτε είμαστε σε καλά χέρια όταν το αναθέτουμε στον Κάρλο. Σημειώνω αυτά τα οποία ελέγχθησαν όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Αλλά αν δούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος, εγώ βλέπω εδώ ένα τεράστιο δυναμικό να ανοίγεται όσον αφορά την καταπολέμηση του εγκλήματος και των εγκληματικών οργανώσεων. Όταν υπάρχει ε, ένα agency, ένας οργανισμός που θα έχει τέτοιου είδους πληροφορίες, όλες αυτές τις βάσεις δεδομένων, που όπως είπε και ο Αλεξάνδερ Άλβαρο, θα μπορούσαν ε, και να συνδυάζονται ως προς τα στοιχεία ε, τα οποία έχουν και να παραπέμπουν η μία στην άλλη. Καταλαβαίνουμε βέβαια τα θέματα προστασίας δεδομένων, αλλά παράλληλα είναι μεγάλη πρόκληση οι δυνατότητες που θα μπορούσε να προσφέρει ένα τέτοιο σύστημα, ένα τέτοιο οργανισμό για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και των εγκληματικών οργανώσεων. Και θα ήθελα να μας πει ο εισηγητής, ενδεχομένως ή και η Επιτροπή, να μας πούν λίγο περισσότερα για αυτή την πλευρά του επιχειρήματος. Επανέρχομαι στον εισηγητή, ο κ. Σκοέλιο. Θα ήθελα να μιλήσω μετά την Κομισιόν και το Συμβούλιο, Πρόεδρε. Άρα δίνω το λόγο στην Επιτροπή, κύριο Στουντοράτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και όλους ε, τους ομιλητές που έθιξαν ε, πολύ σημαντικά θέματα που ήθελα και εγώ να θίξω, όπω είπα, αλλά δεν ήξερα ακριβώ τι σα απασχολούσε και ήθελα να ακούσω τι ερωτήσει για να προσπαθήσω να απαντήσω. Και θα προσπαθήσω να απαντήσω μία-μία τι ερωτήσει και αν ξεχάσω κάτι, παρακαλώ να με διορθώσετε. Προστασία δεδομένων. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα σε κάθε παρέμβαση και είναι σημαντικό να δώσουμε διευκρινήσεις. Ο τρόπος με τον οποίο έχει συνταχθεί τώρα το κείμενο δεν προβλέπει διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων. Επιπλέον, όλοι οι κανόνες που ισχύουν για κάθε ένα από τα συστήματα, και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στην νομική βάση και όλα τα συστήματα που περιλαμβάνουν στοιχεία που έχουν σχέση με την προστασία δεδομένων, όλα παραμένουν διαθέσιμα. δεν αλλάζει κάτι στην πρόσβαση στα δεδομένα ή στο κατά πόσο μπορούμε να, έχουμε, να βλέπουμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα παραμένουν ιδιοκτησία των κρατών μελών. Τα δεδομένα ε, παραμένουν ως κλάστερ ομαδοποιημένα σε κάθε ένα από τα συστήματα. Δηλαδή, ακόμη και αν τα διαχειρίζεται αυτός ο νέος οργανισμός, δεν ε, θα ομαδοποιούνται αυτά τα δεδομένα, που είναι κάτι το οποίο έχει αναφερθεί και στα μέσα ενημέρωσης. Γι' αυτό κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Ε, στο μέλλον δεν ξέρω αν θα υπάρχει μια τάση και επιθυμία να συνδεθούν αυτές οι βάσεις δεδομένων ή να, υπάρξει, να υπάρξουν παράμετροι διαλειτουργικότητας, αλλά και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε πολιτική εντολή. Και αυτό απαντά και τα ερωτήματα για τα μελλοντικά συστήματα. Στον τομέα, στον χώρο ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη, δεν θα προσθεθούν νέα συστήματα στο μέλλον χωρί νέα νομική βάση. Και νομική βάση σημαίνει πολιτική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Και αυτό ο νέο οργανισμό, αυτό καθεαυτό, δεν θα μπορεί από μόνο του ε, να δημιουργεί νέα θέματα, ε, ούτε στον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, ούτε σχετικά με την πρόσβαση των δεδομένων, με τα άτομα που θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, ούτε θα μπορεί να προσθέσει νέα συστήματα ή ε, να ε, δίδει ε, νέο, νέο λειτουργικό χαρακτήρα σε αυτά τα συστήματα. Περιμένουμε και τα σχόλια τα οποία θα λάβουμε από τον επόπτη προστασίας δεδομένων και βεβαίως θα εξετάσουμε και τα δικά σας σχόλια και αν τα θέματα προστασία δεδομένων πρέπει να τονιστούν ιδιαίτερα μέσα στο κείμενο, είμαστε ανοιχτοί να εξετάσουμε ό,τι δυνατότητα υπάρχει. Νομίζω να κάλυψα το θέμα της προστασίας δεδομένων, αλλά αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις που παρέλειψα, ευχαρίστω να τα εξετάσουμε. Τώρα για το θέμα της, του τόπου εγκατάστασης του οργανισμού που έθιξαν κάποιοι βουλευτές. Η Επιτροπή από την αρχή, από τότε που υπέβαλε αυτή την πρόταση, προσπαθεί να κρατήσει μια ουδέτερη στάση. Και το ίδιο το κείμενο ακολουθεί μια ουδέτερη στάση ως προς το θέμα της έδρας, γιατί είναι πολιτική απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί στο κατάλληλο επίπεδο. Όμως, τονίζουμε ότι θα πρέπει να ληφθεί πολιτική απόφαση για τον τόπο εγκατάστασης όσο δυνατόν συντομότερο, διότι το κόστος ε, και οι επιπτώσεις ε, της έδρας ε, στην προετοιμασία και εγκατάσταση του οργανισμού θα είναι σημαντικό. Μπορεί να υπάρξει μία έδρα για το τεχνικό και για το διοικητικό κομμάτι ή μπορεί να υπάρξει και διαχωρισμένη έδρα για τα δύο τμήματα. Όλα αυτά έχουν επιπτώσει στο κόστο. Το αν θα πρέπει να μετακινηθούν τα συστήματα που τώρα βρίσκονται στη Γαλλία και στην Αυστρία, αν θα πρέπει να μετακινηθούν σε άλλο κράτο μέλο, και αυτό επιφέρει κάποιο κόστο. Επομένω, η απόφαση για την έδρα είναι κάτι που μα ενδιαφέρει άμεσα και είναι και σημαντικό στοιχείο στην προετοιμασία αυτού του νέου οργανισμού. Ταυτόχρονα είναι κάτι στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει ουδέτερη. Αναφέρθηκε και το θέμα του προσωπικού. Σας παραπέμπω στην εκτίμηση επιπτώσεων μιλάμε για 120 άτομα ως προσωπικό, εκ των οποίων τα δύο τρίτα θα ασχολούνται με την λειτουργία του συστήματος και το 1 τρίτο θα είναι διοικητικό προσωπικό. Θα είναι ε, σε μεγάλο βαθμό προσωπικό που θα ασχολείται με την τεχνική δουλειά που εξασφαλίζει το σύστημα και στον πρώτο χρόνο μετά την αρχή λειτουργίας του οργανισμού που θα είναι το 2011 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, πρόθεσή μας είναι να προσληφθούν 75 μέλη του προσωπικού, ούτω ώστε να ξεκινήσει η κατάρτισή τους και η προετοιμασία τους για να αναλάβουν τα συστήματα. Ακόμη έγινε μία ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της πρότασης αυτής και του ε, πώς σχετίζεται με τη θέση σε λειτουργία των συστημάτων, ιδίως ε, λόγω των καθυστερήσεων που μέχρι τώρα ε, έχουν υπάρξει για το σύστημα SIS. Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε τώρα κατά νου είναι ότι νομικά θα θεσπιστεί αυτός ο οργανισμός το 2011 και θα αρχίσει να λειτουργεί από το 2012. Εδώ θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ο οργανισμός αυτός δεν αφορά μόνο το SIS αλλά και το VIS και το Eurodac η Eurodac είναι ήδη απόλυτα σε επιχειρησιακό στάδιο. Δεν θέλω να προδικάσω αν θα είναι το πρώτο σύστημα, πάντως σίγουρα αυτό το σύστημα είναι έτοιμο να το αναλάβει ο καινούριος οργανισμός. Και το VIS, ε, το οποίο αυτή τη στιγμή ε, προβλέπεται να είναι έτοιμο το 2010, θα είναι έτοιμο να το αναλάβει αυτός ο νέος οργανισμός. Παρά τις καθυστερήσεις λοιπόν του συστήματος πληροφοριών Schengen, του SIS, δεν φαίνεται να μας φτάνουν αυτές οι καθυστερήσεις πέραν του 2012. Αυτά που προβλέπει η Επιτροπή δεν, προβλέπει, δεν προβλέπουν να πηγαίνουμε πέρα από το 2011. Πάντως ε, αυτός ο οργανισμός δεν θα επηρεαστεί από τις καθυστερήσεις στο σύστημα SIS. Και όταν θα είναι έτοιμο το, ε, το σύστημα SIS θα το αναλάβει αυτός ο οργανισμός, ε, πράγμα το οποίο θα κάνει παράλληλα και με το σύστημα πληροφοριών και τις θεωρήσεις, το VIS και το Eurodac. Επίσης έγιναν ερωτήσεις, θα έλεγα πιο θεμελιώδεις ερωτήσεις για το αν υπάρχει πραγματικά ανάγκη να έχουμε ένα τέτοιο οργανισμό και ο εισηγητή τόνισε στην αρχή, στην παρουσίασή του, γιατί είναι απαραίτητο ένα τέτοιο οργανισμός. Ε, Καθώ αναφορά αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύουμε ότι είναι απλή η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Καταρχήν, ε, η τρέχουσα βάση αναφορά, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο ε, είναι αποδεκτό. Δηλαδή η Επιτροπή από πλευρά νομική και από πλευρά ανθρωπίνων πόρων δεν είναι σε θέση να λειτουργεί αυτά τα συστήματα και η επιλογή του να, τα, να το χειρίζονται τα συστήματα αυτά τα κράτη-μέλη ε, έχει πολλά ε, αντεπιχειρήματα. Αυτή είναι η επιλογή που ονομάζεται γραμμή αναφοράς ΣΥΝ ε, και νομίζω ότι όλα αυτά δικαιολογούν την ε, ανάγκη δημιουργίας ενός νέου φορέα και σα παραπέμπω στην εκτίμηση επιπτώσεων όπου εξετάζεται το αν είναι προτιμότερο ένας νέος οργανισμός έναντι του να έχουμε την επιλογή των υφισταμένων οργανισμών όπως το Frontex ε, κλπ για τα πιλωτικά προγράμματα και το αν θα δώσουμε λευκή επιταγή μέσω του κειμένου αυτού για τη λειτουργία του νέου οργανισμού, όπως έχει τώρα ο οργανισμός, το άρθρο 6 για τα πιλωτικά προγράμματα, ε, αναφέρει ότι κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη για ένα πιλωτικό πρόγραμμα, ή ένα πιλωτικό σύστημα. Πάντοτε θα γίνεται πολιτική συζήτηση κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει γίνει σχετική συζήτηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν εγκρίνουμε το κείμενο αυτό, διότι και η Επιτροπή δεν ήθελε να έχει ο οργανισμό την ικανότητα να αποφασίζει μόνο του να ξεκινήσει ένα καινούριο σύστημα ή ένα νέο πιλωτικό πρόγραμμα προ την Α ή τη Β κατεύθυνση. Είτε αυτό αφορά νέα λειτουργικά στοιχεία στα υφιστάμενα συστήματα, είτε αυτό αφορά τη δημιουργία νέων συστημάτων. Σαφώς λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί το κείμενο δεν δίνει λευκή επιταγή στον νέο αυτό οργανισμό. Δεν νομίζω να μου διέφυγε κάτι. Νομίζω ότι έχω απαντήσει όλα τα ερωτήματα που είχα σημειώσει. Αλλά αν υπάρχει κάτι που δεν απάντησα, παρακαλώ να μου το επαναλάβετε. Ευχαριστώ πολύ. Now, Mr. Hammerstedt, on behalf of the Swedish... Ο κύριος Χάμερστετ εκ μέρου της Σουηδικής Προεδρίας, αν θέλει το λόγο, πριν ξαναδώσω το μικρόφωνο στον εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία ακούσαμε. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή την προσέγγιση έχουμε κι εμείς έναντι αυτής της προτάσεως. Και εμείς έτσι την ερμηνεύουμε, έτσι την κατανοούμε. Εις ό,τι αφορά την έδρα αυτής της υπηρεσίας, στο κεκτημένο Σέγγεν στην ομάδα εργασίας και εκτιμένου Σέγγεν στους κόλπους του Συμβουλίου γίνεται συζήτηση σύμφωνα με την οποία η έδρα δεν θα πρέπει να αποφασιστεί ή δεν θα πρέπει να προταθεί στην ομάδα μας αλλά σε υψηλότερο κλιμάκιο στους κόλπους του Συμβουλίου και δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει ποια διαδικασία θα ακολουθήσουμε για την υποβολή προτάσεων για την έδρα. Δεν θεωρούμε δε ότι η απόφαση για την έδρα θα ληφθεί κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας, οπότε έχουμε προσεγγίσει την ε, επερχόμενη Ισπανική Προεδρία για να λάβει το θέμα υπόψη της. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω. Ευχαριστώ. Must remind... Να μην ξεχνάμε και την ώρα. Ένα λεπτό κύριε Άλβαρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ένα απλό ερώτημα. Ξέχασα να ρωτήσω κάτι. Εφόσον αυτή η Επιτροπή ασχολείται και με θέματα τρομοκρατίας και γνωρίζουμε πόσο λεπτό είναι το, το ζήτημα αυτό, η υπηρεσία αυτή θα είναι μια από τις λεγόμενες κρίσιμες υποδομές. Δεν βλέπω τίποτα που να λέει στο έγγραφο βάσει δεδομένων που θα αντανακλά αυτό το θέμα αν χαθούν τα δεδομένα αυτά και πέσουν στα λάθος χέρια μπορεί να υπάρξει και πρόβλημα με την ίδια την, ε, με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, μπορούν να αντιγραφούν κάπου αυτά τα δεδομένα. Μπορούμε να κάνουμε μια αποκεντρωτική προσπάθεια Ο εισηγητής. Πρόεδρε, τρία σύντομα σχόλια. Πρώτον, για το θέμα της υπηρεσίας. Γιατί, ρώτησαν κάποιοι συνάδελφοι, να δημιουργηθεί μια υπηρεσία. Η απάντηση είναι απλή. Όπως υπενθύμησε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή τη στιγμή το σύστημα αυτό, το ΣΥΣ2, το διαχειρίζεται ένα κράτος μέλος. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι αυτή η κατάσταση θα πρέπει να τερματιστεί και ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό μέσο. Ένα ευρωπαϊκό μέσο δυνάμει της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι δυνάμει της διαδικασίας της διακυβερνητικής ε, συνεργασίας. Έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Αυτό το κοινοβούλιο απεφάνθη υπέρ της εναλλακτικής δημιουργίας μιας υπηρεσίας αυτή ήταν η σαφή άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια πρόταση που αντιβαίνει αυτή τη δικής μας τοποθέτηση, Μάλλον που ε, δέχεται τη δική μας ε, πρόταση. Οπότε αυτό θα πρέπει να το χαιρετήσουμε. Οπότε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό που είπε ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή, ότι δεν θα υπάρξει σύγχυση των συστημάτων, δεν θα υπάρξει επικοινωνία, συγκοινωνία, επικάλυψε, συγχώνευση αυτών των δεδομένων. Δεν υπάρχει νομική βάση για κάτι τέτοιο και θα ήταν επικίνδυνο και από πλευρά προστασία δεδομένων. Δεν είναι λοιπόν αυτό ο στόχο. Το είπε σαφώ ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Όχι στη διαλειτουργικότητα. Το είπε. Τα δύο συστήματα θα συνεχίσουν να είναι ανεξάρτητα αυτόνομα. Και αυτό το χαιρετίζω ως πολύ θετικό. Τρίτο θέμα. Πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι αν κάτι είναι σαφές αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Αυτό είναι απόλυτα σαφές, είναι κοινό στοιχείο όλων των παρεμβάσεων. Και τέλος, για να ολοκληρώσω, λέγοντας ότι δεν θέλω και εγώ να μπω στην ιστορία της έδρας, διότι είναι ένα πολιτικό ζήτημα όπου το Συμβούλιο βεβαίω έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Και δεν έχω μιλήσει ακόμα και με του σκιώδει εισηγητή. Δεν γνωρίζω λοιπόν την άποψη αυτή τη Επιτροπή Πλήρου και των πολιτικών ομάδων. Την προσωπική μου άποψη λέω για την έδρα. Ότι θεωρώ πλέον λογικό να μην υπάρξει γεωγραφική διάχυση των εδρών. Τι εννοώ να είναι η έδρα εκεί όπου θα είναι και η τεχνική συνιστόσα του συστήματος διαχείρισης των δεδομένων. Άκουσα τον Αλεξάνδρ Αλβαρό και έχει δίκιο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα shadow station, ένα mirror site όπως λέμε. Δηλαδή ένα σημείο όπου θα έχουν αντιγραφεί αυτά τα δεδομένα για περίπτωση ο Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ το πρόσθετο ερώτημα του κυρίου Άλβαρο μπορεί να απαντηθεί γραπτώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν συμφωνεί ο εκπρόσωπος αυτής. Ας ακούσουμε πρώτα τον κύριο Λουί Μισελ που ζήτησε το λόγο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Να μην ξανανοίξουμε τη συζήτηση. Όχι, όχι πρόεδρε καθόλου. Δεν θέλω να ξανανοίξω τη συζήτηση. Ένα ερώτημα αφελές έχω. Δεν βλέπω ποια είναι η προστιθέμενη αξία δεν λέω ότι είμαι υπέρ αυτού. Λέω, δεν βλέπω ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτή τη υπηρεσία από πλευρά αποτελεσματικότητα αν δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα. Α μου εξηγήσει τη ποια είναι η προστιθέμενη αξία. Ποιο είναι το νόημα δημιουργία μια νέα υπηρεσία χωρί να υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων. Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Αν είναι δηλαδή να ασχολούνται με αυτά τα συστήματα οι διάφορε εθνικέ υπηρεσίε, δεν βλέπω την προστιθέμενη αξία. Λοιπόν, εγώ μόνο με τη διατηρητικότητα βλέπω ότι να έχει νόημα δημιουργία Δεν λέω ότι είμαι υπέρ αυτού, ούτε και σώνει, έτσι. Απλώ μια απορία εκφράζω. Δεν επίστην δηλαδή από αυτά που άκουσα για τα εκτέλεση των επιχειρημάτων ε, που δεν ήταν καταληκτικά, που δεν ήταν πιστικά ε, και για τις ε, δαπάνες, πέρα από τη δαπάνη δηλαδή και το κόστος. Και επαναλαμβάνω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα καθόλου ούτε για τη χρησιμότητα της υπηρεσίας, αλλά ούτε και για τα λοιπά θέματα. Και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Κοέλιο, προς Θεού ας μην κατακαιρματίσουμε τις διάφορες ε, υπηρεσίες ε, και να μην ξέρει η αριστερά τι πει η δεξιά. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ να απαντήσω σε αυτό το πολύ κέριο πιστεύω ερώτημα. Το backup system προβλέπεται. Θα συνεχίσει να υπάρχει λοιπόν, υπάρχει ήδη, προβλέπεται με την έννοια ότι υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει όταν, συνεχί... όταν ξεκινήσει τις εργασίες η υπηρεσία. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για τη σαφήνεια και την λακωνικότητά σα. Κύριε Κοέλιο, ένα καταληκτικό σχόλιο. Ουχή. Καλώ. Σα ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση προς το παρόν. Ready to continue as we proceed to point number number 13, Σημείο 13. Δημόσια πρόσβαση στο Κοινοβούλιο, στα έγγραφα του Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Θα ακούσουμε πρώτα τον εισηγητή, τον κύριο Μάικλ Κάσμεν και μετά θα δώσουμε το λόγο, θα δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου και μετά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μάικλ Κάλσμαν, παρακαλώ. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ που ξαναγυρνάμε στο πάρα πολύ σημαντικό αυτό θέμα χαιρετήσω τα νέα μέλη στο ζήτημα αυτό γιατί εγώ από το 99 μόλις τέλειωσε το σχολείο άρχισα να ασχολούμαι με το θέμα αυτό ε, έχω περάσει τόσο χρόνο ασχολούμενος με το θέμα αυτό που πρέπει να πάρω σύνταξη όπου να είναι. Τέλο πάντων, και λέω στην Επιτροπή Παρεπιτώντο ότι μην περιμένει να συνταξιοδοτηθώ, θα συνεχίσω να ασχολούμαι. Είναι πολύ σημαντική η πρόταση αυτή που συζητούμε σήμερα. Το Μάρτιο όταν την πρωτοείδαμε αποφασίσαμε να μην κλείσουμε την πρώτη μας ε, αναγνωσή ούτως ώστε να μπορέσει το Κοινοβουλίο να έχει περισσότερες δυνατότητες να αρχίσει άτυπες ε, διαπραγματεύσεις δηλαδή το Κοινοβούλιο με τα άλλα δύο θεσμικά όργανα και να μην δέσουμε αν θέλετε τα χέρια μας στη στιγμή, λίγο πριν από τις ευρωεκλογέ, πριν από το τέλος της θητείας. Τέλος πάντων εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, το Κοινοβούλιο λέει ότι ο κανονισμός που εφαρμόζεται πρέπει να, θεωρεί, να αναθεωρηθεί, να γίνουν κάποιες αλλαγές. Έγιναν κάποιες αλλαγές, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από την ομολογία του ΔΕΚ σε πάρα πολλές υποθέσεις, π.χ. στην υπόθεση Τέρκο για τα των... και στην υπόθεση Λάγκερ. Να πω και κάτι τι άλλο. Η Κομισιόν βέβαια δεν συμφωνεί μαζί μου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πίστευε ότι αντί να πάμε ένα βήμα μπροστά και να αυξήσουμε τη διαφάνεια με, με αυτά που προτείνονται εδώ πίσω γυρίζουμε και η διαφάνεια δεν βελτιώνεται. Το Κοινοβούλιο ε, αποφάσισε ότι, λοιπόν ότι τα πράγματα ήταν έτσι και ο τότε υπουργό, ε, ο τότε πρόεδρος του Κοινοβουλίου έστειλε στα άλλα θεσμικά όργανα μια επιστολή λέγοντας ότι δεν έγινε πλήρης αναδιατύπωση, δεν έγινε σωστά και γι' αυτό συνεχίζουμε να συζητούμε την πρόταση αυτή. Αρνηθήκαμε λοιπόν να κλείσουμε την πρώτη ανάγνωση, έτσι να κάνουμε την τελική ψηφοφορία για την πρώτη ανάγνωση. Και εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και την Επιτροπή που συνεργάστηκε μαζί μου, αλλά πραγματικά ε, έχουμε, είμαστε σε ένα σημείο που επιγόντως πρέπει να προχωρήσουμε. Οι νομικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής ε, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητήσαμε να ασχοληθούν και πάλι με το θέμα γιατί πιστεύουμε ότι εδώ υπάρχουν αντιφάσεις και πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, γιατί θέλουμε να τα δει αυτά η νομική υπηρεσία. Η πολιτική θέση του Κοινοβουλίου είναι δεδομένη ε, εκτός μιας τροπολογίας οι υπόλοιπε τροπολογίες είναι σύμμορφες με τη συνθήκη μια ε, τροπολογία μόνο για μια τροπολογία μόνο δεν συμφωνούμε το Συμβούλιο και η Κομισιόν και πάλι καλά διότι διαφορετικά να μην ερχόμαστε καν εδώ καθόμαστε σπίτι μας η όλη υπόθεση κυρίες και κύριοι είναι σχετικά με το με τη διαφάνεια και τη δημοκρατία. Ε, κάποιοι από τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στις ε, τροπολογίες του Κοινοβουλίου αναφέρονται ακριβώς αυτό και φαντάζομαι ότι θα ότι συνάδουν και με την ορολογία της συνθήκης Λισαβόνας αλλά θα υπάρχει ένα κενό και δι κυρίως νομικό τι θα γίνει με όλες αυτές τις agencies, τους οργανισμούς τις υπηρεσίες, τα γραφεία τα οποία δημιουργήθηκαν και τα οποία πρέπει και αυτά να είναι διαφανή, ανοιχτά και δημοκρατικά και εδώ νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα άρθρο 255 της ε, ε, συνθήκης τι θα γίνει με το Europol, με το Eurojust με την προστασία των δεδομένων διότι τώρα μπαίνουμε στα χωράφια του τρίτου πυλώνα ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, που συνδέονται με όλα αυτά τα θέματα πώς θα τα επιβάλλουμε γι' αυτό σήμερα θα ήθελα πραγματικά να κουβεντιάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να καλύψουμε αυτό το νομικό κενό και αυτό το θεωρώ επίγον η δική μου πρόταση είναι τριμερής διάλογος σε πολύ ψηλό επίπεδο για να ξαναδούμε την αναθεώρηση αυτή του 1049 επιγόντως και να γίνει και μια άτυπη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών για τη συζήτηση αυτών των θεμάτων. Νομίζω ότι όλοι θα ενημερωθούν ακόμη και δεν το ξέρουν για την ιστορία της όλης αυτής της υπόθεσης μέσω των γραμματιών τους. Αυτά εν είδη εισαγωγή. Αυτή είναι η πρόταση που κάνω για το αύριο και, αλλά θα ήθελα να ακούσω και από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή την άποψή τους. Η, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως και αυτή βρίσκεται σε ένα κενό. Είναι έτσι rather πόρτε, ε, όπως ο Γκράτσο Μάρξ, δεν ξέρω είδατε εκείνο το, το έργο που λέει ότι α, ωραία, σαν περιστρεφόμενη πόρτα είναι και οι αρχές μου, άμα δεν μου αρέσει κάτι, τι πάω παρακάτω, ε, δε, προχωρώ παρακάτω και πάω στο επόμενο. Ε, αυτά λοιπόν νομίζω ότι και η Κομισιόν βρίσκεται σε ένα κενό. Ευχαριστώ πολύ. Και ας ακούσουμε την κυρία Χίλμπεργκ εκ μέρους της Προεδρίας του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ που καλέσατε τη Σουηδική Προεδρία στη συνεδρία της Επιτροπής σας. Και στο παρελθόν είχαμε ιδιαίτερα επικοδομητική συνεργασία με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για το θέμα αυτό και με τον ίδιο εισηγητή και με μεγάλη χαρά περιμένουμε τη συνεργασία μας και αυτή τη φορά. Η διαφάνεια, όπως και το 2001, αποτελεί προτεραιότητα για τη Σουηδική Προεδρία και η δημόσια πρόσβαση ε, και η πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα επίσης ε, ε, είναι ένα θέμα προτεραιότητας για μας. Σχετικά με τις εργασίες μας στο Συμβούλιο, θέλω να σας πω ότι έχουμε κάνει μια λεπτομερή εξέταση ανάρθρο, μόλις ολοκληρώθηκε και σε αυτή την εξέταση ανάρθρο συζητήσαμε και κάποιες από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Μάρτιο, όχι όλες τις τροπολογίες σας όμως. Στο Συμβούλιο συμφωνούμε με κάποιες προτάσεις της Επιτροπής σας, αλλά όχι με όλες. Δεν έχουμε ακόμη μια τελική προσέγγιση, αλλά έχουμε μια εικόνα των θέσεων των κρατών μελών για τα διάφορα θέματα. Στην ομάδα εργασία ε, του Συμβουλίου αποφασίσαμε να αναβάλουμε τις περαιτέρω συζητήσεις για την πρόταση της Επιτροπής μέχρι ότου ακούσουμε και τον προγραμματισμό του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Περιμένουμε λοιπόν ε, τα νέα στοιχεία, αλλά στο μεταξύ η Σουηδική Προεδρία είναι πρόθυμη να συζητήσει μαζί σας το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον κανονισμό 1049, πώς να βελτιώσουμε τη διαφάνεια και να ενισχύσουμε τα δικαιώματα του κοινού για πρόσβαση στα έγγραφα. Και ιδίως ε, εν ώψη της συνθήκης της Λισαβόνας. Περιμένουμε την τελική επικύρωση και θα θέλαμε να ακούσουμε και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως σχετικές τροπολογίες μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε τώρα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον κύριο Κάσμαν. Και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κάσμαν ε, που ε, επανεξελέγει. Νομίζω ότι όσοι έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό το θέμα πολλά χρόνια τώρα, ε, χαιρόμαστε που συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας από κοινού και ο κύριο Κάσμαν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεργαστεί και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο για να προχωρήσει αυτό το θέμα. Σα συγχαίρουμε λοιπόν και πάλι και περιμένουμε με χαρά τη συνεργασία μα κατά του προσεχεί μήνε. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απολύτω με την ανάλυση του κύριου Κάσμαν σχετικά με τη συνθήκη της Λισαβόνας που όλοι ελπίζουμε ότι θα τεθεί σε ισχύ σύντομα μετά το πολύ επιτυχημένο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία. Η νέα συνθήκη αφορά σε μεγάλο βαθμό τον ανοιχτό χαρακτήρα, την απλούστευση, τη δημοκρατία και τη σαφήνεια. Και στην αίθουσα αυτή σήμερα αρκετοί από εμά ε, ήμασταν και στην συνέλευση και στη διακυβερνητική διάσκεψη όπου συντάχθηκαν κάποια αυτά τα άρθρα και θυμόμαστε τι συζητήσει που έγιναν για τη διατύπωση αυτών των άρθρων, των άρθρων και αντικατοπτρίζεται το πνεύμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο βασικό στόχο τη Επιτροπή και βάσει τη συνθήκη τη Νίκαια ε, παραμένει, δηλαδή θέλουμε να έχουμε μια Ευρωπαϊκή ε, Ένωση ανοιχτή και διαφανή για του πολίτε. Και είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό, διότι όταν μιλάμε για πρόσβαση στα έγγραφα, μιλάμε για πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, πρόσβαση των πολιτών. Δεν θα πρέπει να συγχαίρεται αυτό με το πώ λειτουργούν τα θεσμικά όργανα μεταξύ τους και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία τώρα που έχουμε και το νέο κοινοβούλιο σύντομα θα έχουμε και τη νέα ευρωπαϊκή επιτροπή και με βάση και τη νέα συνθήκη θα δουλέψουμε και με τις μελλοντικέ ε, προεδρίες. Το πώς συνεργάζονται τα θεσμικά όργανα είναι διαφορετικό θέμα. Εδώ μιλάμε όμως ε, ε, για το δικαίωμα του κοινού να έχει πρόσβαση στα έγγραφα. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Και αν έχουμε θέματα τα οποία θέλουμε να ρυθμίσουμε μεταξύ μα, υπάρχουν οι διοργανικέ συμφωνίε που επίση προβλέπονται στη νέα συνθήκη. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερον, Πριν από 17-18 μήνες, τον Απρίλιο του 2008, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τις επανειλημμένες θέσεις του προηγουμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για το πώς θα χρησιμοποιούμε την αναδιατύπωση ως νομοθετικό μέσο, ε, και αυτό είναι μια κοινή μας φιλοδοξία, γιατί και εμείς συμφωνούμε με την άποψη του Κοινοβουλίου. Και βάσει της συμφωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων για το πώς πρέπει να γίνει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε αυτή την πρόταση ως αναδιατύπωση του κανονισμού Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό για τους πολίτες να μπορούν να διαβάσουν και να κατανοούν το κοινοτικό δίκαιο και είναι πολύ σημαντικό μέσα σε ένα τέτοιο κανονισμό όπως ο 1049 να κωδικοποιούμε το δίκαιο όπως ε, εξελίσσεται. Δεν να γίνει σύγχυση των ε, διαφόρων ε, μέσων. Εμείς πιστεύουμε ότι ακολουθήσαμε το σωστό δρόμο και το κάναμε και βάσει των ε, όσων είχε εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ψηφίσματα και σε επιστολές και στις διοργανικές συμφωνίες μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ένα στοιχείο που θεωρούμε σημαντικό είναι το πώς λειτουργήσε ο κανονισμός 1049 Ε, δεν μιλάμε για την περίοδο ακριβώς μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκη της Νίκης. Ε, δεν μιλάμε για ε, νέο κανονισμό για πρόσβαση στα έγγραφα. Έχουμε κανονισμό για πρόσβαση στα έγγραφα και τώρα έχουμε και 8 χρόνια πείρας πάνω στη δουλειά με ένα τέτοιο κανονισμό. Και σε αυτό το διάστημα και εσείς στο Κοινοβούλιο και εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οι φίλοι μας στο Συμβούλιο έχουμε τώρα μια μακρά πείρα για το πώς λειτουργεί αυτός ο κανονισμός που αποτελεί κατά κοινή ομολογία ένα ε, επιτυχημένο κανονισμό. Όπως θα δείτε και από την ετήσια έκθεση που δημοσιεύουμε, υπάρχουν πολλά αιτήματα προς την Επιτροπή και αυτό είναι λογικό το να έχει η Επιτροπή μεγαλύτερα ε, να έχει περισσότερα αιτήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ε, αντιπροσωπεύουμε μεγαλύτερο όγκο εγγράφων και καλύπτονται στο 80-85% στο άρθρο 4 και εσείς ως νομοθετικό όργανο ε, αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους μπορεί να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα έγγραφα. Η Επιτροπή παραδείγματο χάρη ε, σε σχέση με τον ανταγωνισμό έχει την αρμοδιότητα ε, να αντιμετωπίζει συμπράξεις ή καρτέλ στην αγορά. Εδώ έχουμε κάποια νομικά έγγραφα τα οποία δεν μπορούν να είναι ανοιχτά σε πρόσβαση του κοινού γιατί αυτό θα υπονόμευε το ρόλο της Επιτροπής και αυτό δεν το αμφισβητεί κανένα ούτε το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το έχει αμφισβητήσει. Είναι πολύ επιτυχημένος λοιπόν αυτός ο κανονισμός, ο 1049. Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου και συμφώνησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, θεωρήσαμε ότι καλό θα ήταν να γίνει αναδιατύπωση αυτού του κανονισμού και να συμπεριλάβουμε ε, και ε, νέες ε, εξελίξεις στην νομοθεσία και νέα θέματα τα οποία θα χρειαστεί να λάβουμε υπόψη. Μετά τη συζήτηση που έγινε και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά την δική σας ψηφοφορία του Μαρτίου και μετά τις συζητήσεις που ακολούθησαν στο Συμβούλιο η Επιτροπή συνεχώς εξηγεί τους λόγους για τους οποίους έχουμε κάνει κάποιες τροποποιήσεις στον κανονισμό. Και πιστεύουμε ότι η πρόταση της Επιτροπής ε, που έχετε ενώπιόν σας είναι η σωστή πρόταση και μπορεί να αποτελέσει τη βάση των συζητήσεων. Εμείς υπερασπίζουμε την πρότασή μας γιατί θεωρούμε ότι παρουσιάζει ακριβώς τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν, την κωδικοποίηση ε, ε, της νομοθεσίας και την ε, προσπάθεια του να έχουμε νομική σαφήνεια. Έχουμε ακούσει τα αντίθετα επιχειρήματα και από την αρχή είπαμε ότι με χαρά μας θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και με εσάς και με το Συμβούλιο. Ε, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να θεωρείτε ότι κάποια τροποποίησή μας ε, είναι διατυπωμένες με τρόπο που δεν συμφωνείτε είτε εσείς το Συμβούλιο και ευχαρίστω να αναζητήσουμε τη λύση στις συζητήσεις και με εσά και με το Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε ότι υπάρχει κατανόηση για τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε πρόθυμοι να βρούμε το σωστό τρόπο για να διατυπώσουμε σωστά αυτές τις τροποποιήσεις. Επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η πρόταση της Επιτροπής, ω έχει τώρα, αποτελεί ένα μικρό αλλά καθόλου αμεληταίο βήμα υπέρ της διαφάνειας, μεγαλύτερης διαφάνειας για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφιστώ την προσοχή σας σε μια τροπολογία που το καθιστά υποχρεωτικό για τα θεσμικά όργανα ε, να παρέχουν πρόσβαση στα ε, έγγραφα κατά τη διάρκεια της θέσπισης της κοινωτικής νομοθεσίας ε, στο βαθμό που είναι δυνατό θα πρέπει να ε, καταστήσουμε διαθέσιμα αυτά τα έγγραφα θέλουμε να είναι διαθέσιμα προ το κοινό. Διακόπτει ο πρόεδρο. Παρακαλώ, ε, συγγνώμη σα διακόπτω, αλλά θα πρέπει ε, να συντομεύσουμε τη συζήτησή μα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έκλεινα την παρέμβασή μου τόσο αλλω λέει ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Θεωρούμε ότι ε, συνεχίζει να είναι σωστή αυτή η πρόταση αυτή. Για τα θέματα που έχει θίξει ο εισηγητή σα για τι συνθήκε Λισαβόνα, θέλω να πω ότι διεξάγεται προπαρασκευαστική δουλειά στην Επιτροπή με την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου Κοινοβουλίου για τις απαραίτητες νομικές προσαρμογές που θα χρειαστούν άμεσα μετά τη θέση σε ισχύ της νέας συνθήκης είναι η διαδικασία Omnibus ε, που έχετε ε, δει και στο παρελθόν όταν τίθεται σε εφαρμογή μια νέα συνθήκη και ε, ευχαρίστω να εξετάσουμε μαζί σας αν υπάρχουν κάποια τμήματα και άλλα τμήματα του άρθρου 15 που θα πρέπει να συζητηθούν μεταξύ των θεσμικών οργάνων για να γίνει περισσότερο διαφανής η δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Now, Ερωτήσεις παρακαλώ και έχετε κατά ότι έχουμε πρόβλημα χρόνου και πρέπει να είστε σύντομοι. Κυρία Σόμερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχει δίκιο ο εισηγητή. Έχουν αλλάξει πολλοί βουλευτέ στο νέο κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας. Ίσως έχουμε και μεγαλύτερο ποσοστό νέων μελών. Μπορεί να είμαστε πολύ καινούργοι στο Κοινοβούλιο και καινούργοι στην Επιτροπή. Έχουμε κατανοήσει όμως πόσο δύσκολο είναι αυτό το θέμα, πόσο δύσκολο απέβει στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Και πρέπει να ομολογήσω ότι δεν είμαι εξοικειωμένη με αυτό το θέμα, που δεν ήμουν μέλος της Επιτροπής στην προηγούμενη θητεία. Συμφωνούμε με το θέμα της ε, διαφάνειας. Είναι μια γενική αρχή με την οποία συμφωνούμε. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα και το τόνισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοκρατικό δικαίωμα για την πρόσβαση στα έγγραφα ε, το ερώτημα είναι, και ακριβώς αυτό ήταν και το θέμα της συζήτησης ε, μέχρι τώρα για αυτό το θέμα, πόσο, θα πρέπει να, πόσο μακριά θα πρέπει να φτάσει αυτό το δικαίωμα. Ε, πού τελειώνει η διαφάνεια και πού αρχίζει η προστασία των δεδομένων. Και σήμερα ήδη συζητήσαμε πολύ το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Τι γίνεται με την προστασία λοιπόν αυτών των δεδομένων. Είχα την ευκαιρία να εξετάσω εν συντομία αυτή την έκθεση Ε, και είδα στο κείμενο στο άρθρο 6 παραδείγματο χάριν ε, βλέπω ότι θα μπορούσε να ερμηνευθεί ε, ότι θα μπορούσαν να δημοσιεύονται τα πρακτικά κάθε συνεδριάσεως νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτή καθ' μια τέτοια διάταξη ε, δεν θέλουμε ε, ούτε να αυξήσουμε τη γραφειοκρατία ούτε το κόστος το οποίο θα αντιπροσωπεύει κάτι τέτοιο. οι συνεδριάσεις παραδείγματος χάρη ε, των εθνικών αντιπροσωπιών ε, θα πρέπει ε, να διαθέτουν τα πρακτικά τους και τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης ακόμη και τεχνικών συνεδριάσεων θα πρέπει να είναι ανοιχτές προς το κοινό οι επιστολές οι οποίες αποστέλλονται προς οποιοδήποτε παραλήπτη ή ακόμη και τα μηνύματα ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου και αυτά θα πρέπει να είναι προς δημοσίευση το άρθρο 6, ε, αν το ερμηνεύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, μου δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Ίσως η διατύπωση είναι πάρα πολύ γενική και ίσως ε, θα έπρεπε να γίνει πιο συγκεκριμένη η διατύπωση αυτού του άρθρου. Ε, μετά στο άρθρο 7 που μιλάει και για τα κράτη-μέλη. Αυτό το άρθρο 7 φαίνεται σαν να έρει δικαιώματα από τα εθνικά κοινοβούλια. Θα αποφασίσουμε εμείς εδώ ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα διαθέτουν όλα τα έγγραφά τους ε, προς το κοινό και αν δεν ε, δημοσιοποιούν ε, ένα έγγραφο θα πρέπει να αιτιολογούν έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί δεν δημοσιοποιούν κάποιο έγγραφο. ποιος θα αποφασίζει για το αν θα δημοσιοποιείται ή όχι ένα τέτοιο έγγραφο. Ίσως να μην είναι απόλυτα σωστή η δική μου κατανόηση του κειμένου. Αλλά διαβάζοντάς το αυτά τα προβλήματα διαπιστώνω. Στο κοινοβούλιο μας έχουμε κατά το ίμιση νέα μέλη, άρα είναι ένα καινούριο κοινοβούλιο κάθε φορά μετά από τις εκλογές και γι' αυτό θα πρέπει να τίθενται εκ νέου κάποια βασικά ερωτήματα. Μήπως αυτό το κοινοβούλιο, το νέο κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την πρώτη ανάγνωση, γιατί πρόκειται για κανονισμό, για ένα νομικό κείμενο. Δεν είναι γνωμοδότηση απλώς του Κοινοβουλίου. θα πρέπει να συνεχίσουμε με τη δεύτερη ανάγνωση ε, επί τη βάση της κοινή θέση ε, του Συμβουλίου. Θα μπορούσαμε να υποβάλουμε ε, τροποποιήσεις. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε τώρα με βάση τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν από την προηγούμενη θητεία στην πρώτη ανάγνωση. Μετά από τις εκλογές λοιπόν νομίζω ότι δεν είναι επαρκώς ικανοποιητική αυτή η κατάσταση για το νέο κοινοβούλιο. Μας δίνει τη δυνατότητα ο κανονισμός. Το άρθρο 59 παραδείγματο χάρη ε, λέει ότι ένα νέο νεοεκλεγέν κοινοβούλιο μπορεί ε, να επαναλάβει μια διαδικασία πρώτης ανάγνωσης. Θα ήθελα να ακούσω τη θέση του εισηγητού αλλά και τη θέση της Προεδρίας του Συμβουλίου επ' αυτού. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε μια θεμητή επανεξέταση του κειμένου από το νέο Κοινοβούλιο. Θα μας απασχολήσει πολύ αυτό το θέμα στο νέο Κοινοβούλιο. Και κάτι ακόμη για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν έχει τεθεί σε ισχύ ακόμη. Ναι, μεν απάντησαν ναι η Ιρλανδία, αλλά υπάρχει ακόμη και το θέμα της Τσεχίας. Και θα δούμε αν ε, και στην Αγγλία υπάρχει κάποιο ζήτημα Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, πριν τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, πρέπει να περάσουμε στη δεύτερη ανάγνωση για να αποφασίσουμε πάνω σε ένα τέτοιο θέμα. Ή μήπως θα ήταν προτιμότερο να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θα ήθελα κάποια απάντηση από τον εισηγητή για το θέμα αυτό. Πάντως ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εισηγητή και για την προθυμία του να συνεργαστεί με τους σκιώδεις ε, εισηγητές όπως μας είπε. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και για τους Ευρωπαίους πολίτες και για το Κοινοβούλιο και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και για τα Εθνικά Κοινοβούλια και για τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα γενικότερα και ζητώ την κατανόησή σα γιατί θα πρέπει να φύγω τώρα γιατί έχω μια σημαντική συνάντηση στην αντιπροσωπεία μου. Αλλά θα παραμείνουν οι συνεργάτε μου και θα παρακολουθούν λεπτομερώ τι συζητήσει. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χαουτάλα. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο. Είμαι η ε, σκιώδη συγγετρία από τους Πράσινους σε σχέση με τον κύριο Κάσμαν βέβαια θα ήθελα στον κύριο Κάσμαν θα ήθελα να πω ότι έχω κάποια σχέση με το θέμα γιατί την προηγούμενη ζωή μου ασχολιόμουν με, ασχολήθηκα με την υπόθεση και το 2001 καταφέραμε να πάρθει μια κάποια απόφαση. Υπήρχαν βέβαια κάποια λαθάκια, οι ορισμοί δεν α, ε, α, ε, ήταν ίσως τόσο σαφείς, αλλά το πάρθηκε μια απόφαση και έκτοτε το 10 εξέδωσε και κάποιες αποφάσεις ε, οι οποίες επιβεβαίωσαν ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, Κανείς μας κύριε Κάσμα δεν θα ήθελε να γυρίσει την πατρίδα του λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γυρίζει στα θέματα αυτά. Η Κομισιόν λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι κάνει μια πρόταση η οποία δεν ε, κωδικοποιεί απλώς, δεν αναδιατυπώνει αλλά ε, προσπαθεί να τροποποιήσει όλα ορισμένα πράγματα. Το ΔΕΚ ίσως δεν θα ήταν σύμφωνο όσον αφορά τη διαδικασία με αυτά που ε, προτείνει τώρα η Κομισιόν. Θεωρώ ότι έγινε ήδη κάποια δουλειά στην πρόταση της Κομισιόν αλλά βεβαίως υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν ε, και νομίζω κύριε Κάσμαν ότι βρίσκεστε στο σωστό δρόμο Είστε έτσι κι αλλιώς σε επαφή με τη Σουηδική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα θέλαμε πράγματι να ε, φροντίστε να ξεκαθαριστούν ορισμένα πράγματα και στην νομοδότηση. Και η κυρία Σάμερ θα ήθελα νομίζω να ε, είναι βέβαιη ότι οι εθνικές αντιπροσωπείες δεν πρόκειται να κατασκοπεύονται αν θέλετε όσον αφορά τα πρακτικά τους τα, τα, θεσμικά όργανα ακολούθησαν τα τελευταία χρόνια του κανονισμό αυτό για τα δικά τους τα έγγραφα και από εκεί και πέρα βεβαίω έχουμε και τι νομικέ υπηρεσίε, οι οποίε ασχολούνται με κάποια σημεία και περιμένουμε τι απαντήσει του. Θα ήθελα τώρα πέρα από αυτά να θέσω και εγώ κάποιε ερωτήσει. Η Επιτροπή πώ. Ε, η Κομισιόν τι λέει, λέει ότι ουσιαστικά νομοθετικές πράξεις είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συζητήθηκαν μέσα στις ε, διαδικασίες συναπόφαση και τα λοιπά. Στη Φινλανδία ο ορισμός της νομοθεσίας είναι διαφορετικές βάσει του συντάγματός μας. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προσέξει. Πρόεδρος, ε, την προσοχή σα του γεγονός ότι καθυστερούμε. Έχουμε καθυστερήσει. Ε, ο κύριος Δεγιόν και μετά η νομική υπηρεσία της, ε, του, της Κομισιόν. Ευχαριστώ πρόεδρε, λέει ο κύριος Δεγιόν. Νομίζω ότι είναι πράγματι σημαντικό το ζήτημα αυτό. Στις ευρωεκλογέ είδαμε ότι υπήρχε ένα έλλειμμα εμπιστοσύνη από πλευράς πολιτών. Γιατί, διότι η διαδικασία λήψη αποφάσεων στα διάφορα θεσμικά όργανα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ουσιαστικά μαύρο κουτί για τους πολίτες και βεβαίως ε, είμαι καινούριο και στην Επιτροπή αυτή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν θα προσπαθήσω να ανατρέψω τα υφιστάμενα αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε με ένα καινούριο μάτι ε, ορισμένα πράγματα δεν συμφωνώ με την ε, κυρία Σόμερ που λέει ότι θα πρέπει να γίνει πιο περιοριστή θα γίνει πιο περιοριστική περιοριστικές οι διατάξεις εδώ όχι λιγότερο περιοριστικές πρέπει να γίνουν και έχει δίκιο ο κύριος Κάσμαν που είπε το ίδιο πράγμα την πρόταση η δική μου η ομάδα πιστεύει ότι αν ο κανονισμός λέει ότι θα πρέπει να υποβάλλονται αιτήματα πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένα αυτό δημιουργεί πρόβλημα η πρόσβαση στις πληροφορίες ε, για να έχει κανείς πρόσβαση κάποιες πληροφορίες ως πολίτες θα πρέπει να ε, μπορώ να να, να είναι εύκολη για τον πολίτη. Δεν λέω ε, ο πολίτη δεν πρέπει να έρθει να πει θέλω να ξέρω συγκεκριμένα το τάδε η τάδε νομοθετική πράξη τι λέει, αλλά να πει θέλω να ξέρω τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή. Έτσι, ε, λοιπόν, νομίζω ότι δεν μπορούμε να είμαστε πιο περιοριστικοί. Ε, πρέπει να είμαστε να, προσέξουμε και εγώ από πλευρά ε, σας υπόσχομαι ότι θα προσέξω να ανοίξω αυτό το μαύρο κουτί που δημιουργείται εδώ από την πρόταση Πρόεδρος η νομική υπηρεσία μήπως θέλει να πει κάτι τι, διότι έχουν τεθεί διάφορα θέματα και εγώ έστειλα επιστολή με συγκεκριμένα ερωτήματα στην ε, νομική υπηρεσία. Ο κύριος Μπερίλο θέλει να μου απαντήσει. Ναι, Πρόεδρε, πρώτα-πρώτα να επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο Μάικλ Κάσμαν στην αρχή της εισαγωγή που έκανε. Και εγώ όταν ήμουνα πιτσίρικας στο δημοτικό Θυμάμαι ότι στην είσοδο του σχολείου έλεγε η διαφάνεια είναι διαφάνεια είναι δημοκρατία. Υπογραφή Μάικλ Κάσμαν. Λοιπόν, ο κύριο Κάσμαν ασχολείται πολύ καιρό με όλα αυτά τα πράγματα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί του μα είπε και μια ιστορία από μια κομμωδία του Γκράτσο Μάρξ ο κύριος Κάσμαν να πω κι εγώ ότι ε, για το πινκ πονγκ που ήταν μεγάλο παίκτη πινκ πονγκ τέλο πάντων ότι ε, ξεκινήσαμε και εμείς το ξεκίνησε ο Μάικλ Κάσου το πινκ πονγκ με τους Αμερικανούς πριν γίνει μεγάλη δύναμη η Κίνα τέλος πάντων δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσουμε όμως όπως λέει ο Μάικλ Κάσμα να ξαναστείλουμε το μπαλάκι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γι' αυτό λέμε ότι άλλα που πρότεινε ο κύριος Κάσμαν, ε, η τριμερής διάλογος σε πολύ ψηλό επίπεδο, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, μπορούμε να το κάνουμε ειδικά για τούτη την αναδιατύπωση των νομοθετικών πράξεων, για αυτόν εδώ τον κανονισμό. Μέχρι εκεί συμφωνούμε. Βέβαια ετέθησαν και άλλα ερωτήματα ενδιαφέροντα πρόεδρε και αναφέρθηκε το ενδεχόμενο να επανυποβληθούν οι τροπολογίες που ήδη ενεκρίθησαν το Μάρτιο για να ξαναεγκριθούν και να ξανά γίνει πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Συγγνώμη, πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου δεν έχει τυπικά γίνει, δεν έχει υπάρξει σχετική ψηφοφορία. Απλώς ε, νεκρίθησαν όλες οι τροπολογίες και η Επιτροπή πήρε θέση για αυτές τις τροπολογίες. Νομίζω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να ξαναεγκριθεί καμία πρώτη ανάγνωση που έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, δεν ανακρίθη ποτέ. Άρα το μπαλάκι δεν ξαναγυρνάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο διότι δεν υπήρξε ποτέ πρώτη ανάγνωση. Η νομική υπηρεσία τώρα θα ε, μου απαντήσει στην επιστολή που στείλατε πρόεδρε και ευχαριστούμε. Να ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Κάσμαν τότε λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που πήραν το λόγο και είναι κρίμα που έφυγε η κυρία Σόμνερ γιατί η κυρία Σόμνερ έκανε την ε, μεγαλύτερη παρέμβαση. Θα ήθελα να την καθισχάσω πρώτα πρώτα και ε, εκείνη και τον κύριο Μπουστήλ σας καθισχάσω μονίμως αυτός ο σκοπός της ζωής μου κύριε Μπουστήλ. Λοιπόν, για τη συνθήκη της Λισαβόνας, μην πιστεύετε τον κίτρινο τύπο που διαβάζετε και τα κουτσομπολιά στους διαδρόμους. Ο... Άμα γίνει η κύρος και επικύρωση της συνθήκης της συγγνώμη, οποιασδήποτε νομοθετικής πράξης, τότε παρα... είναι νομοθετική πράξη αυτό το πράγμα και αν και εφόσον ε, το ίδιο πράγμα θα γίνει με τη συνθήκη της Λισαβόνας και για να ξεγίνει αυτό χρειάζονται μεγάλες διαδικασίες λοιπόν να αφήσουμε κατά μέρος το Ηνωμένο Βασίλειο και τι φαντάζεται ορισμένοι ότι μπορεί να γίνει λοιπόν Τώρα για το φίλο της νομικής υπηρεσίας να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά που είπε, ιδιαίτερα για το άτομό μου. Εγώ εκείνο που θέλω να γίνει είναι να γίνει μια συνάντηση και σκιωδών εισηγητών και η παραπληροφόρηση ουσιαστικά που έγινε από την Επιτροπή θα συνεχιστεί νομίζω. Εγώ συνεχίζω το πινκ πονγκ. Ή, ή τα προβλήματα των άρθρων 6 και 7 ε, άλλοι λένε ότι δεν είναι εύκολο εγώ νομίζω ότι δεν πειράζει πάει το μπαλάκι πέρα δόθε και από εκεί και πέρα για το την Ολομέλεια το Νοέμβρη ας ε, θέσουμε το θέμα να δούμε τι θα γίνει. Η απα... απάντηση θα πάρετε στην επιστολή σας πρόεδρε. Εδώ μπορεί να διχαστεί το σώμα, αυτό είναι γεγονός, αλλά τι να κάνουμε, that's life. Λοιπόν, και νομίζω ότι ε, θα πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας και να μην ε, λιποψυχήσουμε. Ωραία λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ πλήρως με αυτά που είπε ο συνάδελφος Κάσμαν. Πρέπει να ζητηθούν, είναι θεμελιώδες, διευκρινήσεις στην νομική υπηρεσία ό,τι αφορά τις συνέπειες της συνθήκης Λαφρανώνας επ' αυτού του φακέλου και νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία όλα τα όργανα και υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμορφωθούν με την επιταγή της διαφανείας. Σήμερα, ίσως περισσότερο παρά ποτέ, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να πισωγυρίζει, δεν μπορεί να κάνει πισωγυρίσματα. Έχουμε αναλάβει δέσμευση να προστατεύσουμε αυτά τα δικαιώματα και να υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη διαφάνεια όχι μόνο για τις ε, γνωμοδοτήσεις, για τις ψηφοφορίες αλλά ε, και κυρίως θα έλεγα για τις διεθνείς συμφωνίες όπως η ACTA, SWIFT ή ακόμα και ε, να δώσουμε δικαίωμα πρόσβασης στα πρακτικά διαπραγματεύσεων ας πούμε ε, που είναι τρέχουσες όπως αυτή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λιβύης ο κύριος Μπεσούτιλ ευχαριστώ ευχαριστώ πολύ τον Μάικλ που μου λέει ότι ο σκοπός της ζωής του είναι να μην καθησυχάζει με καθησυχάζει, που σκοπός του ζωή του είναι να με καθησυχάζει. Αν υπάρχουν παρανοήσεις για το πώς θα πρέπει να κινηθούν τα πράγματα, θα πρέπει να αρθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Επί τη βάση λοιπόν αυτής της διαπίστωσης και με την ε, στιβαρή καθοδήγηση του Μάικλ και των σκιωδών, ε, εισηγητών νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια διέξοδο. Άλλα σχόλια πριν κάνει τα καταληκτικά του σχόλια ο εισηγητής. Όχι. Κύριε Κάσμαν. Θέλω να επαναλάβω, Πρόεδρε, αυτό που είπα προηγουμένως. Θα συνεργαστώ με όλους, συμπεριλαμβανομένων και των σκιωδών εισηγητών. Και θα τα λάβω υπόψη μου αυτά στο νέο κείμενο το οποίο θα υποβάλω τον Νοέμβριο στην Ολομέλεια, όπω επίση θα λάβω υπόψη μου βεβαίω και τη γνωμοδότηση τη νομική υπηρεσία. Μάλιστα, λέγει ο Πρόεδρο. Συμφωνούμε λοιπόν. επί της ε, μεθόδου που ανέφερε ο κύριος Κάσμαν με την συζήτηση με τους σκιώδεις εισηγητές και την ε, γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Συνεχίζουμε λοιπόν με το επόμενο σημείο το 14 για τον κατάλογο των τρίτων χωρών των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων. Είχαμε μια πολύ έντονη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα. Η, η αποφάσισε να μεταβεί στο Σαράγεβο την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή και είμαι σίγουρος ότι μπορεί τώρα να μας φωτίσει με τα σχόλιά τη και τι παρατηρήσει τη πριν δώσω το λόγο στους εκπροσώπους της Επιτροπή και του Συμβουλίου. Παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση όταν εκλήθηκε στην Επιτροπή ΑΦΟ η Σάρα Λάτφορντ ετοίμασε μια σχετική γνωμοδότηση. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Η ψηφορία ήταν 51 ψήφοι υπέρ. Πολύ καλό αποτέλεσμα. Θέμα που εντάσσεται στην απελευθέρωση της υποχρέωσης της για τα Δυτικά Βαλκάνια. Πιστεύω ότι η συμφωνία θα είναι καλή, όπως θα προκύψει στην Ολομέλεια εγώ προτείνω η Βοσνία, και η Αλβανία ήδη τώρα προσωρινά να μπουν στον λευκό κατάλογο Σέγγεν αλλά να αρθούν υποχρεώσεις θεώρησης μόνον όταν και οι δύο χώρες ε, πληρώσουν τις ε, υποχρεώσεις τους δυνάμει του συγκριτικού πίνακος επίδοσης. Τώρα, για την επίσκεψή μου στο Σαράγεβο την περασμένη εβδομάδα, πολύ χρήσιμη πολύ ενδιαφέρουσα. Είχα δύο ημέρες συζητήσεων με πολλούς εκπροσώπους της κυβερνήσεως οι οποίοι με ενημέρωσαν πλήρως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ε, στο 90% των υφισταμένων των εκκρεμόντων benchmarks όπως λέμε για να συνεννοούμαστε και έχουν την πλήρη υποστήριξη των πολιτών της Βοσνίας και Ζεγοβίνης. Τον Ιούλιο η Κομισιόν είχε, α, δεν είχε συμπεριλάβει την Βοσνία Ζεγοβίνη στην διαδικασία αυτή, κάτι το οποίο την έθεσε σε ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση. Μετά την επισκεψή μου στο Σαράγεβο μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ήδη πολύ δύσκολη πολιτική κατάσταση θα επιδεινωθεί αν δεν αποστείλουμε ένα θετικό και ισχυρό πολιτικό μήνυμα προς τις αρχές ότι έχει γίνει ουσιαστική και σημαντική πρόοδος για την καταπολέμηση της διαφθοράς, του ξεπλήματος χρήματος, της χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Ε, έχουν υπογράψει και συμφωνία για την ανταλλαγή των αστυνομικών δεδομένων. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η έκδοση των βιομετρικών διαβατηρίων που είχε καθυστερήσει, αλλά <clears throat> δεν ε, αναμένονται προβλήματα θα εκδώσουν γύρω στα 65.000 βιομετρικά διαβατήρια μέχρι το πέρας του έτους. Ακόμα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα παραδέχθηκε όταν ήμουν στο Σαράγεβο ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να αποστείλουμε πλέον αυτό το ισχυρό πολιτικό μήνυμα προς τις ε, αρχές της χώρας ότι τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να τους θέσουμε προσωρινά στον λευκό κατάλογο και όταν πληρώσουν τα εκκρεμή benchmarks θα προχωρήσουμε σε νέα αναθεωρήση της στάσης μας. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω κάποια σχόλια για το Κόσοβο. Είναι λεπτό Βεβαίως το ζήτημα και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις διάφορες θέσεις, τις διαφορετικές θέσεις που εκπροσωπούν τα διάφορα κρατημέλη. Προσπαθούμε λοιπόν σε συνεργασία και με τους δύο σκιώδεις εισηγητές να βρούμε μια συμφωνία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ νέου για την συνεργασία. Εις ό,τι αφορά το Κόσοβο θα ήθελα να πω ότι είναι το μόνο κομμάτι των Δυτικών Βαλκανίων που είναι πλήρως εκτός της διαδικασίας απελευθέρωσης υποχρέωσης θεώρησης. Γνωρίζω ότι είναι επίμαχο το ζήτημα, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι θα πρέπει να εξεύρουμε μια λύση για τους κόσοβάρους πολίτες να βρουν ένα τρόπο να συμπεριληφθούν στη διαδικασία απελευθέρωσης τη ε, της υποχρέωσης ε, θεώρησης. Σήμερα το πρωί έλαβα μια επιστολή πολλοί φοιτητέ, νέοι άνθρωποι προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή μαζί μου όταν ήμουν στο Σαράγεβο. Έλαβα πολλέ επιστολέ ε, ενθουσιώδους ε, υποδοχή τη υποστηρίξη που του έδωσα που αποτελεί για αυτούς μια αχτίδα φωτό στο κατά τα άλλα ζωφερό σκηνικό. Γιατί λέγουν ότι λόγω των κλειστών συνόρων ε, τους καταλαβαίνω. Εγώ είμαι από τη Σλοβενία. Δεν έχουμε κλειστά σύνορα πλέον, αλλά είχαμε για αιώνες. Και η επικοινωνία με τις όμορες χώρες είναι τεράστιο πλεονέκτημα. Εμείς το ζήσαμε αυτό. Οπότε ας κάνουμε κάτι και για αυτούς τους ανθρώπους, ούτως ώστε να μην απομονωθούν. Ευχαριστώ κυρία Φαγιόν. Ακούσαμε τις προτάσεις σας για την Αλβανία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Yes, please. Uh, yes. Please identify yourself, please. Voilà. Um, alors, de la part de la... Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θέλω να πω ότι υπήρχε μια προθεσμία για, την, ε, για τις χώρες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής ε, του Ιουλίου για τη Βοσνία και την Αλβανία για να υποβάλουν συμπληρωματική έκθεση ώστε να εξετάσουμε την πρόοδο στο πλαίσιο της διαδικασίας απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίου. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι όντως λάβαμε πριν από λίγες μέρες, στις αρχές Οκτωβρίου, την έκθεση της Βοσνίας και της Αλβανίας για τις προόδους ε, στο πλαίσιο απελευθέρωσης του καθεστώτος θεώρησης διαβατηρίου. Διαπιστώνουμε με ικανοποίησή μας ε, την πρόοδο που υπάρχει. Επιβεβαιώνουμε αυτό που διαπίστωσε η κυρία Φαγιόν. Υπάρχουν πρόοδοι για τις μεταρρυθμίσεις και για το κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια που αναγράφονται στον χάρτη πορείας και αξιολογούμε αυτή τη στιγμή τις πρόοδους που αναφέρθηκαν. Πολλέ φορέ συμπεριλαμβάνονται μέτρα τα οποία ελήφθησαν την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, παραδείγματο χάρη. Και η αξιολόγησή μας καλύπτει όχι μόνο την έγκριση μέτρων, αλλά και την πραγματική υλοποίηση των μέτρων. Σύμφωνα με την παρακολούθηση της Επιτροπής μέχρι τώρα, Ε, χαίρομαι διότι είχαμε και την ε, υποστήριξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα ε, πριν από λίγο πήραμε την επιβεβαίωση ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο. Τα μέτρα λοιπόν τα οποία ελήφθησαν τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να τα παρακολουθήσουμε για να δούμε κατά πόσο θα υλοποιηθούν στην πράξη και θα οριστικοποιήσουμε την αξιολόγηση των εκθέσεων που λάβαμε πριν από τρεις-τέσσερις μέρες και θα κάνουμε και επιτόπου αποστολές αξιολόγησης σχετικά με τη Βοσνία και την Αλβανία αυτά. Επίσης θέλω να πω ότι λάβαμε και έκθεση από το Μαυροβούνιο και την Σερβία και όπως σας είχα πει πριν από λίγες μέρες, προβλέπονται αποστολές επιτόπου για την επόμενη εβδομάδα στην Κορίτσα και στο Βελιγράδι και στα διοικητικά σύνορα με το Κωσυχοπαίδιο. Σας έχουμε αναγγείλει αυτές τις αποστολές αξιολόγησης, θα τις κάνουμε την επόμενη εβδομάδα και θα προσπαθήσουμε ε, να επαληθεύσουμε το αν πληρούνται τα κριτήρια τα οποία απέμεναν για τις δύο αυτές χώρες. Και η πρόθεσή μας είναι αρχές Νοεμβρίου να υποβάλουμε μια έκθεση για τα αποτελέσματα αυτής της συμπληρωματικής αξιολόγησης που θα γίνει για το Μαυροβούνιο και τη Σερβία την επόμενη εβδομάδα. Αυτά είχα να σας πω και ευχαρίστω να σας απαντήσω σε ερωτήσεις που τυχόν έχετε. Ευχαριστώ κυρία Κόγου. Έχω ένα κατάλογο ομιλητών και παρακαλώ να κρατήσετε το χρόνο να είστε σύντομοι. Κυρία Κοράτσαβιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω κοιόδηση εισηγήτρια, συμφωνώ με την συνάδελφο και φίλη Τάνια και χαιρετίζουμε την πρόοδο η οποία επετεύχθη ιδίω στη Βοσνία πρόσφατα. Και εγώ τις τελευταίες μέρες ε, ήρθα σε επαφή με γνωστούς και με τον υψηλό εκπρόσωπο στην Βοσνία και με την Επιτροπή και βλέπω ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα για να τηρήσουν τα κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι όταν επιμένουμε στη θέσπιση κριτηρίων αυτό λειτουργεί στην πράξη και έχει αποτελέσματα. Η προσέγγιση μας, θέλω να πω, είναι κοινή γιατί όλοι θέλουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία χορήγησης ε, θεώρησης διαβατηρίου σε αυτούς τους πολίτες ε, των χωρών ε, της Βοσνίας, της Αλβανίας, του Μαυροβουνίου και της Σερβίας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Η διαφορά μας με την έκθεση της εισηγητρίας είναι ότι θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί με αυτούς τους πολίτες και να μην τους κοροϊδεύουμε. Θα τους πούμε ότι είστε ευπρόσδεκτοι όταν είστε έτοιμοι. Η διαφορά μεταξύ παρατήματος 1 και 2 είναι νομικό θέμα και όχι πολιτικό, σε όποιο καθεστώς και αν βρίσκεσαι. Δεν μπορεί να είσαι σε δύο παρατήματα ταυτόχρονα, δεν μπορεί να είσαι στο θετικό παράρτημα με αστερίσκο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι προς τους πολίτες. Θα τους πούμε ότι είστε ευπρόσδεκτοι, σχεδόν έχετε μπει. Μόλις ολοκληρώσουμε τη διαδικασία θα είστε κι εσείς μέσα σε αυτό το σύστημα με τους ίδιους κανόνες όπως και όλοι οι άλλοι. Θέλουμε όμως να είμαστε ρεαλιστές και αυτή είναι η δεύτερη διαφορά μας με την εισηγήτρια. Θέλουμε να υποβάλουμε στο Συμβούλιο μια πρόταση που θα είναι αποδεκτή γιατί ξέρουμε ότι το Συμβούλιο δεν θα αποδεχτεί μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Συμβούλιο στην Επιτροπή, πράγμα το οποίο προτείνει η συγγήτρια. Από τη στιγμή που υποβάλλει θετική έκθεση η Επιτροπή, αυτόματα, χωρίς ε, άλλο κανονισμό του Συμβουλίου, να χορηγούνται θεωρήσει διαβατήριο. Αυτό, όπως το γνωρίζουμε, δεν είναι δυνατόν. Γιατί να μην επιταχύνουμε λοιπόν τη διαδικασία. Να κάνει η Επιτροπή τη διαδικασία την αξιολόγηση το συντομότερο δυνατόν, να την υποβάλει στο Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν και μόλις πληρούνται τα κριτήρια δεν θα υπάρχει κανένας ε, λόγος ε, αντιδικίας. Εμείς θέλουμε να προχωρήσει γρήγορα μια διαδικασία ομαλή. Αυτός είναι ο σωστός ε, και λογικός τρόπος να φροντίσουμε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνουν το ίδιο μήνυμα προς το λαό της Βοσνίας, Αλβανίας, Μαυροβουνίου, Σερβίας και Φιρόμ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να συνεχίσουμε τον επικοδομητικό διάλογο που είχαμε και με τη Σάρα και με την Τάνια. Ευχαριστώ. Κυρία Γκόντς, ευχαριστώ. Χαίρομαι που, που συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση και θέλω να υπενθυμίσω ότι αυτή η συζήτηση δεν είναι απλά μια τεχνική απόφαση, δεν είναι απλά μια νομική απόφαση, είναι μια υψηλά, υψηλού χαρακτήρα πολιτική απόφαση και συμφωνούμε όλοι από αυτού. Η σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια, πραγματικά όλοι γνωρίζουμε ότι είναι προ όφελο ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο θέμα θεώρηση διαβατηρίου, είναι θέμα συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν ακολουθήσουμε την πρόταση της Τάνια, νομίζω ότι δημιουργούμε μια πολύ αυστηρή διαχωριστική γραμμή μεταξύ αυτών που παίρνουν ε, την ε, απελευθέρωση θεωρήσεων διαβατηρίου και των άλλων δύο που δεν ε, την παίρνουν αυτή τη στιγμή. και από την, την απάντηση της Τάνια που είπε για την επίσκεψή της τις τελευταίες μέρες και ε, ε, μετά την ε, έκθεση της Επιτροπής δεν πρέπει να δημιουργηθεί μια τέτοια διαχωριστική γραμμή. Δεν έχει σωστή βάση μια τέτοια διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ομάδων, γιατί έχουν κάνει μεγάλε πρόοδου ε, ε, και οι άλλε χώρε προ την ε, πλήρωση των κριτηρίων. Και το πολιτικό μήνυμα θα είναι πολύ διαφορετικό αν πούμε ότι τρει χώρε παίρνουν το καθεστώ ελεύθερη χωρί διαβατηρίου και οι άλλε θα πρέπει να περιμένουν. Ή αν πούμε ότι μόλι όντω πληρούν όλα τα κριτήρια κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως το καταλαβαίνω, είναι μια συνεχής διαδικασία. Δεν είναι τρεις χώρες έναντι δύο. Είναι μια συνεχής διαδικασία. Όταν πληρούν τα κριτήρια, μπορούν άμεσα να συμπεριλαμβάνονται στο καθεστώς ε, ελεύθερων θεωρήσεων διαβατηρίου άμεσα. Ε, και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον ενθαρρυντικό χαρακτήρα που θα έχει η απάντησή μας και γι' αυτό τονίζω επανειλημμένα τη σταθερότητα σε αυτή την περιφέρεια. Είναι πολιτική ευθύνη αυτή η οποία έχουμε και γι' αυτό υποστηρίζω την Τάνια και θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν μπορέσουμε να βρούμε μια λύση που να μην εντείνει τη διαχωριστική γραμμή αλλά με κάποιο τρόπο να δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις χώρες ε, να κάνουν μεγαλύτερα βήματα για να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κυρία Λαντφόρντ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι και πολιτική και τεχνική απόφαση το να δώσουμε ε, θεώρηση διαβατηρίων ελεύθερες σε αυτές ε, τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Και δεν θα ήθελα να υπάρχει έλλειψη σαφήνειας, γιατί δεν θέλουμε ε, να μπερδέψουμε τα κριτήρια, ούτε θέλουμε να είναι θολά τα κριτήρια. Υπάρχουν τα θέματα ασφάλειας των συνόρων, επιβολής του νόμου κλπ. Δεν είναι προς συμφέρον κανενός να κάνουμε κάτι τέτοιο ούτε για τις χώρες αυτές ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να είναι καθόλου θολά τα κριτήρια που θα επικρατούν. Αυτό το οποίο αποτελεί πολιτική απόφαση είναι το αν θα στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει εμπόδιο εκτός από την πλήρωση των κριτηρίων. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να στείλουμε ένα τέτοιο μήνυμα. η απόφαση στην Επιτροπή ΑΦΕΤ ε, συμφωνεί με την ε, θέση αυτή. Ήταν 51 ψήφοι έναντι 8. Είναι δηλαδή μια απόφαση εκ μέρους όλων των πολιτικών ομάδων ε, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΛΚ και θα ήθελα αυτό να το τονίσω και προς την κυρία Κράτσαβιλ συμπεριλαμβάνουμε και τις πέντε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε ένα νομικό μέσο, αλλά υπάρχει μια σταδιακή υλοποίηση η οποία εξαρτάται απλά και μόνο από το πότε αυτές οι χώρες και οι κυβερνήσεις τους θα είναι σε θέση να πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις στο βαθμό που να μπορεί η Επιτροπή να πει ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εκφραστεί τελικά επ' αυτού. Όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται διάλογος και αυτό το απευθύνω σε ερώτημα και προ την Προεδρία και προ την Επιτροπή. Μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτό το θέμα Ξέρετε ότι έχουμε δώσει και ένα ρόλο στο Συμβούλιο, αλλά πρέπει να δούμε αν μπορούμε να βρούμε ένα τρόπο να το κάνουμε σωστά. να μην πρέπει να περάσουμε πάλι από μια ολόκληρη νομική διαδικασία για να έχουμε ένα εντελώ νέο νομικό κείμενο την επόμενη χρονιά από την Επιτροπή με διαβούλευση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και να επανέλθουμε μετά στην Επιτροπή. Θα πρέπει να έχουμε ένα ε, νομικό μέσο, μια νομική πράξη, χωρίς να αποδυναμώνουμε όμως τα κριτήρια. οι εν λόγω χώρες είναι αυτές που θα έχουν την ευθύνη και οι πολίτες θα πρέπει να πιέσουν τις χώρες τους ε, ώστε να μπορέσουν να πληρούν τα κριτήρια και να επιτύχουν αυτό που θέλουν. Είναι μια νομική δομή λοιπόν ε, και δεν αποδυναμώνουμε τα κριτήρια με αυτή τη διαδικασία. θέλω να ζητήσω και από τα άλλα δύο θεσμικά όργανα να μα βοηθήσουν. Και αν δεν σα αρέσει η διατύπωσή μα βοηθήστε μα να βρούμε μια καλύτερη διατύπωση για να εκφράζουμε αυτό που θέλουμε. Αλλά νομίζω ότι τίθεται εδώ μια θεμελιώδη ε, επιλογή. Αλλά υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να το επιτύχουμε και δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγχυση από αυτού. Η κυρία Φαγιόν και εγώ συμφωνούμε και με την ψηφοφορία 51 προς 8 η Επιτροπή Αφέτη νομίζω υποστηρίζει ακριβώς αυτή τη θέση του ότι πρέπει να έχουμε ένα νομικό μέσο. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι την Επιτροπή. Πήραν τις εκθέσεις από τη Βοσνία, Ζαγοβίνη και Αλβανία και θα αξιολογήσουν αυτές τις εκθέσεις, μας είπαν. Και είπαν επίσης ότι θα οργανώσουν αποστολές επιτόπου. Πότε θα γίνουν αυτές οι επιτόπιες αποστολές σε μία τροπολογία μου και η Επιτροπή ΑΦΚΟ προτείνει μηνιαίες αξιολογήσεις από την Επιτροπή για τις χώρες που δεν πληρούν άμεσα τα κριτήρια και θα ήταν χρήσιμο αν μπορέσει να αναλάβει δράση η Επιτροπή σχετικά με αυτές τις επιτόπιες αποστολές και γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε πότε θα κάνετε αυτές τις επιτόπιες αποστολές στη Βοσνία, Ζεγοβίνη και Αλβανία. Και επίσης κάτι ακόμη για το κοσυφοπαίδιο. Όπως και η κυρία Φαγιόν. Θέλω και εγώ να πω ότι θέλουμε να έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση για να βρούμε έναν τρόπο για το διάλογο για θεωρήσει διαβατηρίου με το Κωσυφοπαίδιο, ούτω ώστε να έχουμε ένα χάρτη πορεία για την απελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίου. Όλοι γνωρίζουμε βέβαια τι ευαισθησίε που υπάρχουν σε αυτό το θέμα και ε, η διατύπωση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ε, ε, λέει να μην προδικάζεται η αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θα έλεγα να μην προδικάζεται το καθεστώς του κοσυφοπεδίου, γιατί 23 χώρες είναι υπέρ της ανεξαρτησίας και είπαν δεν ισχύει πλέον το καθεστώς του UNSCR, δεν είναι πλέον προτεκτοράτο των Ηνωμένων Εθνών. Πιστεύω ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας βοηθήσει να διατυπώσουμε νομικά σωστά αυτό το σημείο. Ίσως αυτό το οποίο λέω ε, για την ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών να το εκφράσουμε με μια υποσημείωση ή κάτι τέτοιο. Θα ήθελα όμως ε, να μας βοηθήσει η Επιτροπή και από νομικής και από διοικητής πλευράς για να εκφράσουμε αυτό το οποίο θα ήταν σωστό. Η Επιτροπή ΑΦΕΤ ε, ήταν ξεκάθαρη στην απόφασή της και ελπίζω ότι και η κυρία Κράτσαμπίλ θα συμφωνήσει με την ε, πλειοψηφία για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλουμε να ανοίξουμε την πίσω πόρτα για τις θεωρήσεις διαβατηρίου για την Βοσνία, και Αλβανία. Πρέπει να πληρούν τα κριτήρια αλλά δεν χρειάζεται μια νέα νομική πρόταση από την Επιτροπή και να μην επαναλάβουμε την όλη διαδικασία ξανά. Αλλά να προσπαθήσουμε μόλις πληρούν πλέον τα κριτήρια ε, να εφαρμόζεται άμεσα το καθεστώς. η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν κάποιο νομικό, τεχνικό πρόβλημα, γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αυτή τη λύση. Ευχαριστώ. Κύριε Λάντφορντ ε, έχει υποβάλει μια γνωμοδότηση που υπευλήθησε σε ψηφοφορία στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και ξέρουμε ότι είναι ένα από τα πολύ ευαίσθητα θέματα αυτό το θέμα. Αλλά κλείνοντα αυτή την ε, πρωινή μα συνεδρίαση θα πρέπει να έχουμε κατά νου το χρόνο που μας απειλεί και μέχρι τις 12.30 πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Γι' αυτό σας παρακαλώ να κρατήσετε το χρόνο σας. Η κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ. Ω και όδη της ομάδας μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρία Φαγιόν Είμαι από την Ανατολική Γερμανία και βεβαίως και κατανοώ πόσο σημαντική είναι αυτή η πρόταση την οποία μας έχετε διατυπώσει και πόσο σημαντικό είναι για μια περιφέρεια να τελειώσει τον κύκλο απομόνωσης ε, και να κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση όχι μόνο για την Αλβανία και την Βοσνία Ζεγοβίνη, αλλά θα πρέπει να ανοίξουμε και στο κοσυφοπέδιο τη δυνατότητα. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή διατύπωση για να μην ανοιχτεί μια τέτοια επιλογή. Και παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τη θέση της και να λάβει υπόψη στη θέση και των άλλων ε, χωρών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί προς αυτή την ε, έναρξη της διαδικασίας και για το κοσυφοπαίδιο. Είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες που ζουν ε, στις χώρες αυτές και θα είναι σημαντικό να δοθεί ένα μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο προς την κατεύθυνση του ανοίγματο. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει και την πολιτική κατάσταση αλλά και θα δώσει μια νέα όθηση και θα ενθαρρύνει αυτές τις χώρες. Παρακαλώ λοιπόν δώστε ένα τέτοιο μήνυμα για το άνοιγμα του διαλόγου με το κοσφοπέδιο. Πρέπει να χρησιμοποιούμε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται και εγώ θα ήμουν πρόθυμη να εξετάσουμε οποιαδήποτε διατύπωση δίνει μια τέτοια δυνατότητα προς την κατεύθυνση αυτή. Κυρία Τζάνοκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Συμφωνούμε με την θέση της εισηγήτριας. Το συζητήσαμε και στη συζήτηση που έγινε ε, το Σεπτέμβριο και ως εκπρόσωπος ε, της ομάδος των Πρασίνων θέλω να υπενθυμίσω τη θέση μας για τη χρήση βιομετρικών στοιχείων. και αν δεν ήταν ένα από τα απαιτούμενα δεδομένα, νομίζω η διαδικασία θα ήταν ταχύτερη. Θα υποβάλουμε λοιπόν τις σχετικές τροπολογίες. Ξέρουμε ότι αποτελούμε μειοψηφία. Ήμασταν πλειοψηφία και όταν συζητήθηκε το θέμα της Σερβίας αλλά θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι χρειαζόμαστε μια έγκριση λαμβάνοντας υπόψη και τη θέση μας για τα βιομετρικά δεδομένα. Χαιρετίζουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων πάνω στην γνωμοδότηση της κυρίας Λάντφορτ. Ευχαριστώ. Κύριος Μπόνς. Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφής η θέση της ομάδας μας και θα σας πω το λόγο. Η Βοσνία είναι μια χώρα όπου οι ηγέτες των μουσουλμάνων θέλουν να ενταχθεί η Σαρία στο Σύνταγμα και θα αποτελέσει ένα χώρο που θα είναι καταφύγιο τρομοκρατών. Εμείς θέλουμε να προστατευτούμε έναντι χωρών τέτοιου τύπου. Δεν πρέπει να δοθούν παρεκκλήσεις για τη θεώρηση διαβατηρίου για πολίτες μιας τέτοιας χώρας. Είναι κατά των πολιτιστικών μας αξιών και γι' αυτό θέλουμε να προστατευτούμε και είμαστε κατά αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε ε, μία απόλυτα ορθολογική γραμμή ε, και να ακολουθήσουμε την πρόταση της κυρίας Λάτφορντ. Άκουσα αυτό που είπε και η κυρία Κράτσεβιλ και ε, Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. θέλουμε να έχουμε ίση μεταχείριση, αλλά πώ να είμαστε δίκαιοι όταν οι κροατέ που ζουν στη Βοσνία έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν ελεύθερα, γιατί έχουν ένα μεγάλο, μια μεγάλη γειτονική χώρα, την Κροατία, και τι θα γίνει ε, αν έχουν την ευκαιρία αυτή και οι Βόσνοι και οι Σέρβοι ε, της Βοσνίας δεν θέλουμε να πάρουμε μια απόφαση που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερε εντάσει λόγω τη γραμμή που ακολουθούμε. Το να έχουμε μια λευκή λίστα είναι σωστό, αλλά αν δεν πληρούν τα κριτήρια η Βοσνία ή άλλε χώρε, δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ε, ε, να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Αν πληρούν όμως τα κριτήρια θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν. Είναι σημαντικό αυτό και για την καταπολέμηση της διαφθοράς και η συνεργασία με τι χώρε αυτέ θα πρέπει να συνεχιστεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα υπάρξει απελευθέρωση θεωρήσεων διαβατηρίου δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή υπάρχει ο αλφα τρομοκράτης δεν θα δώσουμε θεωρήσεις διαβατηρίου στους άλλους. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα. Κύριος Βίλτσεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να προσθέσω εγώ κάτι στον ευαίσθητο χαρακτήρα που χαρακτηρίζει αυτή την περιφέρεια, θα μιλήσω μία από τις γλώσσες των χωρών των Βαλκανίων. Οι λαοί αυτοί για αιώνες έζησαν μονιασμένοι. Βεβαίως μετά τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας τα πράγματα άλλαξαν. και τα πράγματα είναι δύσκολα όχι μόνο στο Κόσοβο αλλά και στη Μακεδονία, λέει ο και στην Κροατία και αλλού. Από την άποψη αυτή δεν θα πρέπει να επιφέρουμε περαιτέρω διακριτικές μεταχειρήσεις και προβλήματα. Θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους αυτούς όλους με τον ίδιο τρόπο. Είτε είναι σταθερές οι, οι θεσμοί τους, είτε είναι σταθεροί είτε όχι. Είναι θέμα σεβασμού των τεχνικών κριτηρίων, κυρίως των βιομετρικών διαβατηρίων. Δεν θα πρέπει να έχουμε πολιτική λοιπόν θεώρηση των πραγμάτων, αλλά τεχνική θεώρηση των πραγμάτων. Το Κόσοβο δε, αντίθετα από τις άλλες χώρες, είναι ομοιογενής χώρα. Οι Σέρβοι σχεδόν δεν υπάρχουν. οι Σέρβοι έχουν σερβικό διαβατήριο. Δεν θέλουμε λοιπόν οι Κωσοβάροι για να μπορούν να ταξιδεύουν, να βγουν από τη χώρα τους παράνομα ή να αποκτήσουν διαβατήριο άλλης χώρας. Αυτά νομίζω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ως κριτήρια που θα πρέπει να πρετανεύσουν. Ευχαριστώ. Η κυρία Χολμάγερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Με δύο λόγια μονάχα. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι αυτά που είπε ο κύριος Μπόντες δεν ισχύουν και στις δύο ε, περιπτώσεις πρόκειται για διευκολύνσεις τα κριτήρια θα πρέπει να παραμείνουν και να τηρούνται και στο μέλλον και άμα βάλουμε αστερίσκους στο, όταν βάζουμε ε, αστερίσκους στο παράρτημα 1 και παρόλα αυτά ζητείτε η βίζα τότε καταλαβαίνετε ότι ε, ε, κάτι πρέπει να κάνουμε δεν μπορούμε να δώσουμε παρόλα αυτά τη βίζα σε κάποιες χώρες που δεν πληρούν κριτήρια Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα έχουμε παράτημα 2 και κάποιες χώρες που δεν χρειάζονται, για τις χώρες που δεν χρειάζονται θεώρηση. Αν τώρα επιλέξουμε ορισμένες χώρες από εκεί και βάλουμε αστερίσκο εκεί, που σημαίνει δηλαδή ότι γίνονται παράρτημα 1, αυτό από νομική απόψεως ε, ε, ε, είναι λάθος, διότι είναι σαν να διαλύουμε, να αναιρούμε ουσιαστικά το παράρτημα παράρτημα 1. Εγώ νομίζω ότι το παράρτημα 1 όμως το, το χρειαζόμαστε. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι ουσιαστικά παραπλάνηση γιατί δημιουργούμε την εντύπωση σαν να, δω, σαν να σαν να μην χρειάζεται βίζα για αυτούς τους ανθρώπους αλλά ε, παρόλα αυτά χρειάζεται ε, θεωρώ ότι σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις θέλουμε να μην χρειάζονται θεώρηση αυτές οι δύο χώρες ωραία τότε ας ε, ζητήσουμε την τροποποίηση των παραρτημάτων δεν είναι και τόσο περίπλοκο αυτό το περίπλοκο είναι ότι προσπαθούμε από την πίσω πόρτα να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα στα παραρτήματα. Προ... Πρόεδρος, έχει συζητηθεί εκτενώς το θέμα αυτό. Δίνουμε το λόγο στην εκπρόσωπο της Κομισιόν, κυρία Γκόγκου. Θα είμαι πολύ λακωνική. Καταλαβαίνω πολύ καλά την προσέγγιση κάποιων μελών της Επιτροπής σας που λένε ότι χρειάζεται μια πολιτική απόφαση που να να, να αναφέρεται και στις ανάγκες των συγκεκριμένων περιοχών και χωρών. Συγγνώμη, ε, εμείς κάναμε μια πρόταση. Ποιος λαμβάνει υπόψη αυτές τις ανάγκες ε, στην πρότασή μας μιλάμε για τα Δυτικά Βαλκάνια δεν μιλάμε για άλλες χώρες για άλλες ε, περιοχές που περνάνε από το θετικό κατάλογο στον αρνητικό κτλ δεν υπάρχει άλλη καμία διάταξη που να τροποποιεί τον κανονισμό αυτό εκτός ούτως ή άλλως έτσι ε, έγινε και με τις προηγούμενες προτάσεις κομισιών Προφανώς είμαστε υπέρ της πρότασης αυτή. Προφανώς πρέπει να υπάρχει και μία περιφερειακή προσέγγιση εδώ. Η Κομισιόν ανέκαθεν αυτό έλεγε. Μίλαγε για ολόκληρη την περιφέρεια, για ολόκληρη την περιοχή και ορίστηκαν κάποιες διαδικασίες και απλώς επιβεβαιώνω την αρχική μας πρόθεση. Η πρότασή μας επιβεβαιώνει την πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διατηρήσει αυτή την περιφερειακή ε, προσέγγιση. Από εκεί και πέρα για τα κριτήρια είπαμε επανειλημμένως στις ενδιαφερόμενες χώρες ότι θα πρέπει όλοι να αξιολογηθούν αλλά ο καθένας ξεχωριστά ε, για το αν ε, πληρούν κάποια κριτήρια ή όχι. Και εδώ κλείνω διότι νομίζω ότι τα πράγματα είναι σαφή. Βεβαίω θέλουμε συνεκτική προσέγγιση, περιφερειακή προσέγγιση, αλλά αξιολόγηση της κάθε μιας χώρας ξεχωριστά για τα κριτήρια. Τώρα, το 2001 ε, με τη Ρουμανία υιοθετήθηκε και εφαρμόστηκε προσέγγιση με τον αστερίσκο. Η τελική απόφαση όμως να διαγραφεί ο αστερίσκος ήταν η απόφαση του Συμβουλίου μετά από πρόταση επίσημη την τυπική της Κομισιόν η οποία Κομισιόν όμως είπε ότι είχαν γίνει και πρόοδοι δεν ε, δημοσιεύτηκε έκθεση της Κομισιόν και δεν ήταν αυτό εν πάση που έσβησε τον αστερίσκο παρόλο που η πολιτική βούληση υπήρχε στην Κομισιόν το, η, δια, διαγραφή του αστερίσκου περνάει από το Συμβούλιο ε, λέω λοιπόν εκ μέρους της Κομισιόν ότι υποστηρίζουμε γενικώ την περιφερειακή παρε, ε, προσέγγιση γι' αυτό κάναμε πρόταση και για τα δυτικά Βαλκάνια συλλήβδην. Όμως η αξιολόγηση γίνεται ε, ε, ε, ανά χώρα ανά μία, ανά κάθε χώρα ξεχωρι... κάθε, σε κάθε χώρα ξεχωριστά για να δούμε πώς τηρούνται τα κριτήρια σε αυτή, την κάθε μία χώρα. Λοιπόν, θα πρέπει να προσέξουμε επίσης γιατί ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή μπορεί να δημιουργήσει ένα προηγούμενο για άλλες χώρες στο μέλλον. Τώρα, τι θα κάνει η Κομισιόν. Την επόμενη εβδομάδα θα βγάλει μια ανακοίνωση η οποία θα περιγράφει τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί για το κοσυφοπέδιο διότι όντω το κοσυφοπέδιο είναι μέρος της περιοχής δεν πρέπει να το ξεχνάμε όμως έχει και κάποιες ιδιαιτερότητε στο Κόσοβο τη νομική του, το στάτους του και τα αναγνώριση ε, μερική, όχι πλήρες κλπ. Θα συνεχίσουμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση και απαιτείται ενδεχομένω για το κοσυφοπαίδιο ειδική λύση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του κοσυφοπαιδίου. Πριν δώσω το λόγο για τα καταληκτικά σχόλια στην κυρία Φαϊόν, θα ήθελα να πω ότι είναι έτοιμη προς ε, ψηφοφορία στις 19 Νοεμβρίου στην Ολομέλεια του Στρασβούργου αυτή η έκθεση. Δεν θα ψηφίσουμε σήμερα, αλλά στο Στρασβούργο. Τροπολογίες αύριο μέχρι τις 12 το μεσημέρι. 19 Οκτωβρίου, Πρόεδρε. Οκτωβρίου. Ναι, έκανα λάθος. Ναι, 19 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. είναι συνάδελφοι που έχουν κάποιες ε, συναντήσεις εκτός Βρυξελών, γι' αυτό αναβάλαμε την ε, ψηφοφορία. Τα καταληκτικά μου σχόλια. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχή ε, που διαπιστώνω ευρεία πλειοψηφία υπέρ της γνωμοδότηση που ετοιμάζω και εδώ και στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Με χαρά δε άκουσα και τα λεγόμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι υπέρ της προσέγγισης, της άγουσας που λαμβάνουμε. Ελπίζω και εγώ να βρεθεί η σωστή νομική λύση για το πώς προσωρινά θα προσθέσουμε αυτές τις δύο χώρες στον λευκό κατάλογο, την Βοσνία, Ριζεγοβίνη και την Αλβανία και ελπίζω πραγματικά να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε. Και βεβαίως θα λάβω υπόψη μου και τις τροπολογίες που θα υποβληθούν μέχρι αύριο το μεσημέρι. Να τονίσω απλώς εδώ ότι δεν μειώνουμε τις απαιτήσει μας. Ο δρόμος που οδηγεί στην κατάργηση ή στη διευκόλυνση θεωρήσεων είναι ο ίδιος για όλες τις χώρες. Συμφωνώ με την Κομισιόν επ' αυτού. Δεν θέλουμε όμως να χάσουμε πρόσθετο χρόνο. Δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση τη νομοθεσίας. Διότι αν γίνει αυτό, του χρόνου που θα έχει εκλογές η Βουρζία η Βοσνία Ερζεγοβίνη θα βρεθεί σε ακόμα δυσχερέστερη κατάσταση από την οποία, είναι τώρα με τους ε, ε, Σερβοβόσνιους και τους Κροάτες. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ε, συμφωνία. Τώρα που το έχουν κάνει οι άνθρωποι θα πρέπει να τους αποστείλουμε ένα θετικό μήνυμα για να αποφύγουμε ακόμα μεγαλύτερες ρήξεις και σύγκρουσεις στην περιοχή αυτή στο μέλλον. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε εδώ και θα επανέλθουμε στις 3 το απόγευμα για το πακέτο ασύλου.